Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας πω ότι ο πρόεδρος Αλμπερτίνη δυστυχώς κολλείεται σήμερα παρευρεθεί και ζητεί συγγνώμη γι' αυτό. Ε, σας υποβάλλω την ημερήσια διάταξη, τη γνωρίζετε. Σήμερα το πρωί θα εξετάσουμε πρώτα την πρόταση ψηφίσματος για την Ισλανδία είναι για δεύτερη φορά συζήτηση. Στόχος συζήτησης είναι η εξέταση των τροπολογιών, 20 περίπου τροπολογίες κατατέθηκαν, ξέρω με τους συναδέλφων για την έκθεση αυτή, του κυρίου Κριστιαν Πρέντα. Πού είστε κύριε Πρέντα? Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμανικά. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση στην Επίτροπή μας στις 10 Φεβρουαρίου. Έκτοτε έχουν συμβεί δύο σημαντικά γεγονότα σχετικά με την Ισλανδία. Πρώτον, η συμφωνία ISAVE θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα στις 9 Απριλίου, έτσι αποφάσισε ο πρόεδρος της χώρας. Και λαμβάνοντας υπόψη ε, αυτή την κατάσταση υπέβαλα στη συνέχεια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 10 του κειμένου που είχαμε συζητήσει το Φεβρουάριο και θα σας την αναγνώσω. Η Ισλανδική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία στις 17 Φεβρουαρίου 2011 ε, λαμβάνει υπόψη την ε, απόφαση του Προέδρου της χώρας ε, να ε, υποβληθεί σε δημοψήφισμα η πρόταση αυτή για να τερματιστεί η διαδικασία προσβολής η παραβιάση που ξεκίνησε στις 26 Μαΐου του 2010 από την ΕΖΕΣ. Τελειώνει η παράθεση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσθέσουμε εδώ ότι η Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισλανδών είναι υπέρ της νέας αυτής συμφωνίας. Ε, οπότε και θα υπερψηφίσουν φαντάζομαι στις 9 Απριλίου. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι απέτυχε ο έβδομος γύρος διαπραγματεύσεων να βάγισε Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία, Ισλανδία και Νήσι Φερόε για ε, την κοινή διαχείριση των αποθεμάτων ε, σκόμβρου. Ε, ε, σας παραθέτω και πάλι την αντιστοιχή παράγραφο. θα ρίνουμε την Ισλανδία να διατηρήσει το ταχύ βηματισμό της ε, στις διαπραγματεύσεις με στόχο να έχουμε μια ποσόστοση βιώσιμη στο μέλλον και αηφόρο και ε, αυτή είναι η τροπολογία που έχω καταθέσει προφορική για αυτό το δεύτερο στοιχείο. Υποστηρίζω ε, τις περισσότερες τροπολογίες των συναδέλφων, διότι ε, συμπεριλαμβάνουν πολλά χρήσιμα στοιχεία και τα δέχομαι. Υπάρχουν όμως και τροπολογίες οι οποίες δεν μπορώ να δεχτώ. Παράδειγμα, η παριθμόν 1 Τάρατ και ε, Σαρζεντίνη. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν συνδέεται άμεσα με τις ε, ε, διαπραγματεύσεις προσχώρησης και το δεύτερο τμήμα κάνει αναφορά στην εσωτερική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι δεν θεωρώ ότι έχει καμία σχέση αυτό με το ψήφισμα. Στην τροπολογία παριθμών 2 που έχει υποβάλει ο κύριος Δέβα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να φοβούμαστε ε, ότι ε, θα επιταχυθούν οι διαπραγματεύσεις γιατί έρευνα για την iSave. Είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή της Ερευνητική Επιτροπή η ε, έκθεση που προέκυψε για την κρίση και τη χρηματοπιστωτική και τη τραπεζική που συγκλώνησε τη χώρα το 2008. Ε, είναι αρκετά εμπεριστατωμένη και εκτενής. Έχει μελετηθεί πολύ. Επίση πρέπει να σας πω ότι τώρα η ανάκριση και η έρευνα που γίνεται ε, κατά του πρώην Πρωθυπουργού προχωράει με κανονικούς ρυθμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία υπαριθμών 10 ασχολείται με το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Νομίζω είναι πάρα πολύ πρόημο το στάδιο να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε στη διαδικασία ελέγχου ακόμα, screening, screening συγγνώμη, και δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ιδέα αυτή τη στιγμή να εξαιρεθεί, να αποκλειστεί η Ισλανδία από ε, αυτό το σκέλος του κοινοτικού και εκτιμένου. Και τέλος, ε, απορρίπτω διάφορες τροπολογίες που ζητούν πλήρη ή μερική απάλληψη ε, της αναφοράς της κοινή γνώμης στην Ισλανδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα της ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες ε, τροπολογίες, γιατί ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση της κοινή γνώμης είναι σημαντικό. Νομίζω δεν ασφαλώ όταν λέγω ότι η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτική πτυχή όταν ζητούμε, συζητούμε για την πρόσβαση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν άποψη για αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου προέκυψε ότι 56% των Ισλανδών ε, εμπιστεύονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ μόλις 28% εμπιστεύονται τη δική τους Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Watson. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση που μας παρουσιάζει. Ε, νομίζω πιο μακριά από την Ισλανδία δεν θα μπορούσε να ήταν η γενέτειρα του εισηγητή. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα οι φιλελεύθεροι δεν έχουν καμιά σοβαρή ένσταση για το περιεχόμενο της έκθεσης. Θα υποβάλουμε μια-δύο τροπολογίες για τη διατύπωση. Αλλά καταρχήν υποστηρίζουμε το σχέδιο. Τρία είναι τα βασικά ζητήματα κατά τη γνώμη μας. Πρώτον, η βούληση του λαού του ίδιου της Ισλανδίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιμένουμε την επίσημη έκφανση, απόδειξη της βούλησης αυτής. Δεύτερον, αποζημίωση από τις τράπεζες. Είναι καλή η συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα εμπλεκόμενα μέρη κατά τη γνώμη μας και ομολογουμένως κάποιοι από τις τοπικές αρχές και όσοι διερεύνησαν τις Ισλανδικές τράπεζες ε, θα ήταν ε, προτιμότερο να είχαν μεριμνήσει περισσότερο όταν έκαναν τις επενδύσεις τους και να μην ασχολούνται μόνο με τις ε, αποδόσεις ε, των ε, επενδύσεων. Και όπως είπε και ο εισηγητής, βέβαια υπάρχει μία λεπτομερής έκθεση γι' αυτό και εν γέννη μας ικανοποιεί. Τρίτο θέμα, αλία φαλαινοθυρία συγκεκριμένα. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια και τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να δείξουμε ευαισθησία, ε, διότι είναι μια πατροπαράδοτη Ισλανδική βιομηχανία. Αυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να ε, συμμορφωθούμε με τις απαιτήσει ε, που έχουμε προβλέψει για την ε, περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μία ερώτηση για την παράγραφο 6 θα ήθελα να θέσω στον εισηγητή σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια σχετικά με το ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης για τους διορισμούς δικαστικών αξιωματούχων. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να αντιληφθούμε ποια είναι η φύση αυτής της μικρής χώρας της Ισλανδίας. Όλοι γνωρίζουν τους πάντες στην Ισλανδία και τελικά κάποιος πρέπει να φέρει την πολιτική ευθύνη για τις αποφάσεις ε, που λαμβάνονται. Και γι' αυτό ε, το λόγο, αυτό το σύστημα βάσει του οποίου ε, προσδίδεται ιδιαίτερη ευθύνη στον Υπουργό Δικαιοσύνη, ανεπτύχθη υπέρμετρα και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τους Ισλανδούς και να δούμε αν μετά τη συζήτηση θα προτίθενται να τροποποιήσουν το σύστημα. Όμως αναγνωρίζοντας την ιδιάζουσα ε, φύση αυτή της μικρής κοινότητας, της μικρής ε, χώρας, ε, θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση για αυτά τα χαρακτηριστικά της Ισλανδίας. Ευχαριστούμε κύριε Βότσον, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω αν ε, θα μπορούσε ο εισηγητή και λοιπέ πολιτικέ ομάδε να εξετάσουν ε, με προσοχή και ευμενώ στην τροπολογία ένα των Πρασίνων, βάσει τη οποία ε, υποστηρίζεται η πρωτοβουλία για τα μέσα μαζική ενημέρωση, πρωτοβουλία τη Ισλανδική κυβέρνηση. Έχουν γίνει πολύ ενδιαφέροντα πειράματα και νομικό πώ στην Ισλανδία για να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την ελεύθερη πρόσβαση στι πληροφορίε των ΜΜΕ. Θα μπορούσατε να εξετάσετε λοιπόν αυτή η τροπολογία, ίσως να καταλήξουμε σε μια προφορική, αλλά να διατηρηθεί η ουσία παρακαλώ, ε, η δυνατόν στην τελική έκθεση. Σας ευχαριστούμε κυρία μου. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ο κύριος Φέρν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια προ τον εισηγητή. Είναι εξαιρετική η έκθεση. Είμαι πραγματικό μέλο τη Επιτροπή. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Προπολογισμών και μόνιμο εισηγητή για τη διεύρυνση και γι' αυτό με ενδιαφέρει το ζήτημα. Βασικά πιστεύω πω οι προτάσει σχετικά με το πώ θα χειριστούμε τι τροπολογίε δεν μα δημιουργούν πρόβλημα. Θα ήθελα άλλο ιδιαίτερο να τονίσω την ε, σημασία μια ενδεχόμενη ε, απόρρεψη τροπολογία 17 για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η τροπολογία για το όλο θέμα. Θα επανέλθω. Ε, το Μάιο θα στείλουμε αντιπροσωπή από την Επιτροπή μα. Δεν μπορέσαμε να συντονιστούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν πειράζει γιατί δεν μπορούμε να πάμε το φθινόπωρο. Έχουμε διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό. Άρα πρέπει να πάμε το Μάιο. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι από πλευρά τη Ισλανδία υπάρχει βούληση να βρουν λύσει για τα βασικά του προβλήματα. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό για τα οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ σύνθετα και θα κρίνουμε από την έκβαση και του δημοψηφίσματο πώ θα κινηθούμε. Όμω θα πρέπει να καταδείξουν ότι επιθυμούν να βρεθεί μια λύση για δύσκολα ζητήματα όπω τα αλλιευτικά. Δεν ζητούν ε, βαρεκλήσει, δεν ζητούν ξεχωριστέ ε, ε, μεμονωμένε λύσει. Θέλουν να διαπραγματευτούν. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης μπορεί να είναι μεγάλα του για την Ευρώπη η Ισλανδία. Πέρα από τη στρατηγική σημασία είναι πολύ προηγμένη η κοινωνία τους με αυξημένε γνώσεις για σημαντικά θέματα όπως διαχείριση του θαλασσίου, βίου, ενέργεια, ε, ε, αλία κτλ. Εμείς μπορούμε να μάθουμε από αυτούς για αυτά τα ζητήματα. Όμως, όμως και το είπε και ο κ. Γότσον και άλλοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μοναδική περίπτωση η Ισλανδία, πολύ προηγμένη, πολύ σύγχρονη κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως αυτή η κοινωνία ε, ε υπερασπίζεται τη γλώσσα, την κουλτούρα της, τον τρόπο ζωής της, ε, με τα και άρα εμείς πρέπει να βρούμε ευέλικτες λύσεις. Και υπάρχουν και δύο τομείς που δεν προαναφέρθηκαν, που όμως θα δημιουργήσουν θέματα. Η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη υπάρχουν ναι, επαρχίε στην Ισλανδία που διαφέρουν πάρα πολύ από την κατάσταση που βλέπουμε στο Ρέικιαβεκ, παραδείγματο χάρη. Άρα θα πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί, να βρούμε λύσει και για αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ενημέρωση. Και άρα είναι σοφό να απορριφθεί αυτή η τροπολογία 17 κατά τη γνώμη μα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανένα άλλο συνάδελφο το λόγο, ο εισηγητή μα για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Πάρα πολύ σύντομα μου επιτρέπετε. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 6 που ανέφερε ο κύριος Γότσον, η παράγραφος αυτή είναι θετική. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις προσπάθειες που καταβάλουν οι Ισλανδοί για την ε, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το θέμα των διορισμών ε, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι κάτι που ρώτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Γι' αυτό ψηφίσαμε στην παράγραφο αυτή και σημειώνουμε, μάλλον σημειώνουμε τις προόδους που κάνουν οι Ισλανδικές αρχές ε, διατηρώντας πάντα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πάρα πολύ μικρής κοινότητας που ε, είναι αυτό το κράτος τώρα. Σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Χάουταλα, την πρώτη τροπολογία. Όπως σας είπα προηγουμένως, φρονώ ότι αυτή η πρωτοβουλία για τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση. Και για το δεύτερο, μάλλον το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας του κυρίου Τάραντ και της κυρίας Αρχεντίνη προτείνει να αλλάξει το κεκτημένο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται αυτό, πώς θα το κάνουμε. Ε, κατά τα λοιπά θα μπορούσαμε να δούμε αν με άλλο τρόπο μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμ για τα σχόλιά του. Τώρα σε ό,τι αφορά την τροπολογία 17 που ανέφερε και εκείνος, Κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, να το διαγράψουμε και να απαλληφθεί αυτό που αναφέρει παράγραφος 31. Δεν μπορώ να δεχτώ καθόλου την τροπολογία 17. Ευχαριστώ πολύ. Διαφωνούμε από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ενημερώνω για την ψηφοφορία. Θα γίνει το απόγευμα αφού τελειώσει η ανταλλαγή απόψε με την κυρία Άστον. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πρώτη συζήτηση για την έκθεση πρωτοβουλίας της κυρίας ε, Μουνής. Ο, κόσμος, ε, ο Παγκόσμιος Φορέας και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει στις πολυμερείς οργανώσεις μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. για να βοηθήσουμε την εισηγήτρια να κάνει τις προτάσεις, αναθέσαμε εξωτερική μελέτη. Και πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο εμπειρογνώμονες μας που έκαναν τη μελέτη αυτή, η οποία διανέμεται στην αίθουσα. Ο κύριος Μανουέλ Ντελαρόκα και Βινθέντε Παλάσιο από το ε, Ισπανικό Ίδρυμα Αλτερνατίβα, εναλλακτικέ ε, λύσει. Εναλλακτικέ προτάσει. Παρακαλώ σύντομα να μα παρουσιάζετε τα αποτελέσματα τη έρευνα αυτή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή, τη μελέτη για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολυμερείς οργανώσεις, θα πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και να διερευνήσουμε και το πεδίο δράσης. Η έκθεση αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν είναι πλήρης. Πάντα είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε ερωτήσεις και υποδείξεις από πλευρά σας και προτάσεις. Βασικό στόχος της έκθεσης αυτής ήταν να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεγιστοποιήσει τον ρόλο της σε πολυμερείς οργανώσεις μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για το λόγο αυτό επικεντρωθήκαμε πρώτα στη νομική βάση της συνθήκης της Λισαβόνας μέσω μελέτης των νέων αρμοδιοτήτων ε, της Ένωσης στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τη στιγμή και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλλάζει. Αυτό σημαίνει να αποτυπώσουμε τη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα είναι μεγαλύτερη προβολή της, μεγαλύτερη ισχύ της ε, διεθνώς. Επιλέξαμε λοιπόν κάποιες βασικές πολυμερείς οργανώσεις οργανισμούς, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το G20, το ΝΑΤΟ και τον ΟΑΣΕ που είναι κυρίως οργανισμοί ασφαλείας. Δεν έχουμε ε, την αξίωση να καλύψουμε σε 25 σελίδες όλες τις ε, πολυμερείς διεθνείς οργανώσεις. Επίσης προσπαθήσαμε να ε, προβληματιστούμε για το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δυνατότητες και τις πραγματικές δράσεις στην κοινή εξωτερική δράση. Η βασική θέση και η βασική παραδοχή είναι ότι η πολυμερή συνεργασία δεν ε, πηγαίνει καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της διεθνώς και θα πρέπει η διαδικασία αυτή να θεωρείται ως ε, διαδραστική ε, προσπάθεια, συνεργασία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων αφενός και αφετέρου τον εσωτερικό συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βασικές θέσεις για ενίσχυση του μηχανισμού συντονισμού γιατί υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ των δαρβενιστών και των λεγόμενων λειτουργιστών και θα πρέπει και οι δύο πλευρές να εργάζονται ε, σωστά. Η εξωτερική ε, αντιπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γνωρίζει μια παράδοξη κατάσταση. Από τη Λισαβόνα και μετά έχει μειωθεί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να αυξηθεί. Υπάρχουν και προβλήματα και προσκόμματα που ε, προβάλλουν κάποιες χώρες ε, μέλη και αυτό καταλήγει σε κοινό εκπροσώπηση στις διεθνείς αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναβαθμίσει το σημερινό της καθεστώς σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Ε, αν είναι ε, να γίνει πλήρες μέλος, ας πούμε, ή η συμμετοχή της. Και η Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Άστο, θα πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση τη αυτή για να αναβαθμίσει το ρόλο και την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεκτικέ πολιτικέ εξωτερική δράση, ανθρωπιστική συνεργασία, για παράδειγμα, ε, η αναπτυξιακή εμπόριο, μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και επίση. η βελτίωση τη υπηρεσία εξωτερικής δράσης ως προς το προσωπικό τη δεν θα πρέπει να είναι ποσοτική αλλά ποιοτική. Όχι περισσότερους υπαλλήλου, αλλά ενίσχυση ε, για να ε, είναι ταχύτερη η εκπροσώπηση και η αντίδραση ε, στους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που είναι αργή η δράση μας. Έχουμε και προτάσεις για το Κοινοβούλιο. Παράδειγμα. Χρειαζόμαστε κοινό μηχανισμό συμφωνίας, ένα πρωτόκολλο δράσης, όπως δείχνει η σημερινή κρίση στη Λιβύη και πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ε, δίνει τακτικά συστάσεις μέσω εκθέσεων στην ε, ύπατη εκπρόσωπο. Για τα οικονομικά θα τα πει ο συνάδελφος Ρόκα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι απόλυτη προτεραιότητα να μεταρρυθμιστεί το σύστημα για το Ηνωμένα Έθνη. Ε, για τη Γενική Συνέλευση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα προηγμένο καθεστώς ε, παρατηρητή. Ήδη γίνονται κινήσεις από το περασμένο Σεπτέμβριο και ε, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των λεγόμενων περιφερειακών οργανισμών, περιφερειακής ολοκλήρωσης. να ξεφύγουμε δηλαδή από την εθνοκεντρική λογική που έχει ο Οργανισμός Εθνών, να περάσουμε σε περιφερειακή διάσταση. Δεν ζητάμε μία έδρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βράχει πρόθεσμα, αυτό δεν θα ήταν ρεαλιστικός στόχος, αλλά ζητούμε ε, ε, αύξηση των μονίμων μελών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να υπάρχει υπερενισχυμένη πλειοψηφία για να καταργηθεί το βέτο και να προχωρήσουμε περισσότερο ένα βήμα ε, προς την Ευρώπη της άμυνας, πράγμα που είναι απαραίτητο για την παγκόσμια ασφάλεια. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για την πρόσκληση, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε τον προβληματισμό, τι σκέψει μας και τα αποτελέσματά μας σχετικά με το ρόλο στη διεθνή σκηνή της Ευρωπαϊκής Ένωση. Θα ήθελα, εν συντομία, να σχολιάσω τις συστάσεις μας ε, για τις τρεις οργανώσεις που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Σύνθεση G20. Για το ΔΝΤΑΦ, το Θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ασυνέχεια, διότι έχουμε ένα υπερεθνικό σώμα με παγκόσμια συμφέροντα, ενώ ε, τα μέλη είναι εθνικές οργανώσεις ε, υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την ε, Παγκόσμια Τράπεζα για θέματα όπως ε, η μακροφορολογική πολιτική είναι θέματα μεικτής αρμοδιότητας, αλλά υπάρχει συντονισμός. Ε, πάντως ε, δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση της Ένωσης ούτε με το καθεστώς παρατηρητή. Λοιπόν, για την νομισματική πολιτική στη ζώνη ευρώ δεν υπάρχει φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παγκόσμια Τράπεζα διότι δεν εκπροσωπείται στο εκτελεστικό συμβούλιο ούτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ούτε της Παγκοσμίας Τράπεζας και για τα υπόλοιπα θέματα εστερείται επίσημη εκπροσώπηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου τη Παγκόσμια Τράπεζα, αν βασιστούμε σε εκλογικέ περιφέρειες για τι ψήφου των μικρών χωρών, είναι μία λύση. Δηλαδή, οι πέντε βασικοί μέτοχοι έχουν ε, μεμονωμένε έδρε. Ε, με την εξαίρεση τη Γερμανία, τη Γαλλία και του ΗΠΑ, Βασιλείου, τα λοιπά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται σε ομάδες ε, χωρών που δεν συμπίπτουν όμως ε, με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν και γι' αυτό θεωρούμε ότι με την τωρινή κατάσταση περιορίζεται η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντονίσει τις θέσεις και να λειτουργήσει από κοινού. Οπότε θεωρούμε ότι χρειάζεται τροποποίηση τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να απηχούνται καλύτερα ε, και η διεθνή πραγματικότητα και η διεθνή θέση τη Ένωση. Προτείνουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιζητήσει ε, καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στο εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς Ομισματικού Τμήματο και της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, και να εκπροσωπείται οπωσδήποτε στην Παγκόσμια Τράπεζα όταν είναι θέματα ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητούνται. Ε, χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο για τις, ευρωπαϊκές, ε, ε, για τις χώρες που ανήκουν στη ζώνη ευρώ και έναν πρόεδρο που θα μας εκπροσωπεί στο εκτελεστικό συμβούλιο για τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ. Έχουν γίνει συζητήσεις στο παρελθόν για το θέμα αυτό δεν έχουμε καταλήξει όμως σε μία λύση. Ε, για μία ή δύο ομάδες ε, χωρών ε, θεωρούμε ότι με τη νέα λύση δεν θα μειωθεί η βαρύτητα της ψήφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση των νέων ποσοστώσεων. Τώρα, για το εκτελεστικό συμβούλιο υπάρχει μία συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι G20 τον Οκτώβρη ε, για δύο έδρες κρατών μελών που δεν θα λειτουργούν βάσει του συστήματος εκπεριτροπής, ε, αλλά πρόκειται για δύο μεγάλες οικονομίες. Ε, είναι καλή απόφαση βέβαια γιατί αποφάσισαν να εκχωρήσουν τις θέσεις τους, τάχθηκαν κατά του βέτο και επίσης προώθησαν περαιτέρω τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ε, ως προς τις ποσοστώσεις ε, και τις ε, έδρες να αρχίσει να είναι πλήρω λειτουργικό το σύστημα μέχρι το 2020 με διάμεσο σταθμό το 2010. Το 2012 θεωρούμε μια καλή ημερομηνία ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει η σύσταση Ευρωπαϊκής Εκλογικής Περιφέρειας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας ε, Τράπεζας και μετά το 2020 μπορεί να επιδιώξει μια ε, ενιαία έδρα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. για την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα πράγματα είναι παρεμφερή, όπως και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βασιζόμαστε στα κράτη-μέλη βάσει του συστήματος εκπροσώπησης με εκλογικές ε, περιφέρειες που όμως ε, δεν οδηγεί σε ικανοποιητική εκπροσώπηση των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά ομαδοποιούνται κράτη-μέλη με άλλε χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσωπούνται όλε αυτέ οι χώρε μαζί στο εκτελεστικό συμβούλιο. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία φωνή, ενιαία εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ όμω τα πράγματα περιπλέκονται, διότι οι πολιτικέ ε, δεν είναι αμυγό και κοινοτική αρμοδιότητα, είναι θέματα μεικτή αρμοδιότητα. Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει όμως αρμοδιότητα για την νομισματική πολιτική, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Θα προτείναμε λοιπόν στην περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας το εξή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει μία ενιαία θέση, έδρα διευθυντού στο εκτελεστικό συμβούλιο που θα συμμετάσχει στο μεταρρυθμιστικό ε, πρόγραμμα τη ε, τράπεζα και στην προσχώρηση νέων χωρών, επιδιώκοντα την κατάργηση του βέτο για τη ΣΥΠΑ ε, στο εκτελεστικό συμβούλιο τη Παγκόσμια Τράπεζα. Την ίδια μεταρρύθμιση μπορούμε να εφαρμόσουμε στις πολυμερείς περιφερειακές τράπεζες όπως αυτή της Αφρικής, της Αμερικής, όλες τις περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες. Τώρα, σε σχέση με τη σύνθεση G20 και τη θέση εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέσσερα κράτη-μέλη ανήκουν στο G20, ε, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και προσκαλείται μονίμως και η Ισπανία εκπροσωπείται τριπλά δηλαδή η Ένωση σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο. Σε δύο περιπτώσεις ήταν, συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής G20. Με δύο τρόπους τουλάχιστον μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση της Ένωσης. Πρώτον, οι εκπρόσωποι δεν δηλαδή πρέπει να γίνουν από δύο ένας ε, στις συνόδους του G20. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιος από τους δύο πρόεδρους του Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρευρίσκονται και επίσης θα πρέπει οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες ε, και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής G20 πρέπει να συντονίζουν τις θέσεις τους τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει καλύτερη σχέση, καλύτερο σύνδεσμο μεταξύ του G20 και των Ηνωμένων Εθνών, ε, ούτω ώστε να έχουμε την ομοποίηση των Ηνωμένων Εθνών και στο G20 και προτείνουμε το εξή. Η G20 να είναι ad hoc, ε, ένα ad hoc ε, διυπουργικό εργαλείο που θα συνεργάζεται με το ECOSOC για την εκπόνηση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών ή Ο πρόεδρο ζητά από τον ομιλητή να μιλά πιο αργά. Ναι, αλλά ολοκληρώνω τώρα, πρόεδρε. Η δεύτερη λιγότερο φιλόδοξη λύση, η βραχυπρόθεσμη λύση, είναι οι δύο οργανώσεις, η σύνθεση G20 και τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται χωριστά και όλη η πλήρη νομιμοποίηση των Ηνωμένων Εθνών να μην μετακυλιστεί στο G20, αλλά ε, οι τελικές αποφάσεις G20 και ΠΟΣΟΚ ε, να εξετάζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, να λειτουργούν ως συμβουλευτικοί οργανισμοί δηλαδή, ε, το G20 και το ΕΚΟΣΟΚ. Ε, Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μουνιέθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχει διαφύγει από κανένα και κυρίω στην Επιτροπή μας ότι χρειάζεται παγκόσμια διακυβέρνηση για κοινά προβλήματα και σήμερα αυτή χωλαίνει. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί που λειτουργούν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί τώρα τα θέματα και η περιπλοκότητα τους διεθνώς και μάλιστα ε, με ηλικιώδεις ρυθμούς οι διεθνείς οργανισμοί και τα κράτη βρίσκονται στα όρια της δυνατότητας διαχείρισης αυτών των καταστάσεων. Κινδυνεύουν ορισμένα θεσμικά όργανα, ορισμένοι θεσμοί και οργανισμοί και έχουμε όλο και περισσότερα κλαμπ, λέσχες, επιμέρους ad hoc ε, συνενώσεις κρατών που δεν έχουν πάντα ούτε συνέχεια, ούτε συνοχή, ούτε ε, δημοκρατική νομιμότητα, ούτε υποκαθιστούν τους ε, διεθνείς οργανισμούς. Και επειδή είναι πολύ πολύ πλέον στον κόσμο, χρειάζεται παγκόσμια διακυβέρνηση με στρατηγικό σχέδιο που σήμερα λείπει. Οι παράγοντες κλειδιά έχουν και δυσκολίες με τα ίδια τα εσωτερικά τους ε, σχήματα, όργανα και δομές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν επειδή υπάρχει δυσκολία διαχείρισης κατάστασης και η συνθήκη της φιλοδοξεί ε, να κάνει παγκόσμιο πρωταγωνιστή και πάλι ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μια νέα εξωτερική αρχιτεκτονική. Όλα αυτά ε, συνεισφέρουν έτσι ώστε η έκθεση αυτή και τελικά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς βλέπει το ρόλο του και της Ένωσης διεθνώς είναι πάρα πολύ επίκαιρη και σημαντική συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν θα επιμείνω, έχει ένα σχετικό ειδικό βάρος στον κόσμο παντού και ε, στα εμπορικά θέματα και στο ΕΠ και ε, ως στρατιωτική δύναμη, ως βασικός δωρητής στην αναπτυξιακή βοήθεια, ως ε, συνεισφέρουσα στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ, με πολλά προγράμματα, με πολλές αποστολές και επιπλέον έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας που ε, δίνει μια νέα διάσταση στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή όμως η φιλοδοξία της συνθήκης προσκρούει ε, στη δυσκολία και στις αμφισημίες της ίδιας της συνθήκης. Το σύστημα ε, εκχώρησης αρμοδιοτήτων και η θεσμική πολυπλοκότητα, ο λαβύρινθος αυτός, ιδιαίτερα στην εκπροσώπηση την εξωτερική, είναι πρόβλημα. η διεθνής ε, πρακτική και τα τεκτενόμενα στρέφονται ακόμα γύρω από κράτη ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος. Γι' αυτό ε, προκύπτει μια επιπλέον δυσκολία και χρειάζεται και μεταρρύθμιση της διεθνούς αρχιτεκτονικής για να δούμε πώς θα ενταχθεί ως δομικό συστατικό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, έξω και η εκθεσή μου δεν μπορούσε να είναι γραμμική. Αλλά ε, με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζει τους διάφορους ε, διεθνείς οργανισμούς. Στο σχέδιο αυτό λοιπόν ε, εξετάζω τα προαπαιτούμενα για να δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωταγωνιστής παγκοσμίω μετά την Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι έξι τα μεγάλα κεφάλαια και χωρίζω και σε υποπαραγράφους. Επιλέγω μια σειρά πολυμερών οργανισμών που ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μεγαλύτερη παρουσία. Κάνουμε μια σειρά γενικές ε, συστάσεις αλλά και ειδικέ προς τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή ε, κονίστρα. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν ε, στους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα αναφορά στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, πώς να, το πω, να αντικατοπτρίζει την παγκόσμια συνεργασία, να είναι και ηγητική στην κοινή δράση για τη ε, διακυβέρνηση και για το χειρισμό για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων. Γίνεται λόγος για τη μεταρρύθμιση των διεθνών αυτών οργανισμών επίσης και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επωφεληθεί από αυτές για να ε, ενισχύσει και το δικό της ρόλο και των οργανισμών με στρατηγική εστίαση και κριτήρια ε, συνεκτικά και συνεπής στην εξωτερική εκπροσώπηση με μόνιμη αναθεώρηση των σημερινών ε, συνεννοήσεων και συμφωνιών για την εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να αναβαθμιστεί παντού κατά μία βαθμίδα, κατά μία κλίμακα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί η διεθνής διπλωματία, συλλογική διπλωματία της Ένωσης με τα κράτη-μέλη. Αυτό υπάρχει και στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπαν και εκπρόσωποι εμπειρογνώμονες που έκαναν τη μελέτη, στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία εκπροσώπηση ενιαία, όπως γίνεται στον ΠΟΕ ή στο ΦΑΟ. Ένα αντιπαράδειγμα σε αυτό είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ε, διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, όπου είναι συντρέχουσες αρμοδιότητες αλλά και αποκλειστικές αρμοδιότητες, αλλά δεν μιλάμε με μία φωνή, ε, έχουμε παραφωνία και πολυφωνία. Στις συντρέχουσες αρμοδιότητες επίσης θα πρέπει να έχει ε, μία έδρα η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και από μία ε, τα κράτη-μέλη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Καλούμε προς μία ενίσχυση της θεσμικής ισορροπίας, όπως ακούστηκε, ουσιαστική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Ο κύριος Φερνάντο Γκυμαράες θα μιλήσει νομίζω, είναι παρόν. Ε, στη Γενική Συνέλευση λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών γίνονται ενέργειες για να εγκριθεί ένα ψήφισμα προς την κατεύθυνση αυτή για ουσιαστική πραγματική συμμετοχή διαφορετική από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας στόχος είναι η μεταρρύθμιση του Ήδη με τα τελευταία γεγονότα, αλλά και τα πιο πρόσφατα, αλλά και τα τελευταία χρόνια έχει φανεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσει της παγκόσμιας κοινότητας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να έχουμε συμμετοχή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μάλλον είναι ευσεβής πόθος και πολύ μακράς πνοής. Ε, να υπάρχει όμως συντονισμός και διαβουλεύσεις των κρατών μελών της Ένωσης που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ε, το τρίτο κεφάλαιο αφορά τους διεθνείς οικονομικούς ε, οργανισμούς. Ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου εκπροσώπησε Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τελείως αναποτελεσματική και περιορίζει τη δυνατότητα επιρροής που έχει η Ευρώπη. Παρόλο που έχει και ε, αποκλειστικές αρμοδιότητες σε νομισματικά θέματα, οπότε πρέπει να έχει και μια ε, έδρα στο εκτελεστικό συμβούλιο του Δούνου του. Για την Παγκόσμια Τράπεζα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό ε, το καθεστώς που έχουμε παρατηρητού στο Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να είναι όλα ενωμένα σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια, constituency. Για τον ΟΑΣΕ τώρα ζητούμε καθεστώς παρατηρητού και στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, στο Συμβούλιο Βορειοατλαντικού Συμφωνού για να ε, προσαρμοστούμε στο πνεύμα της Σύνθεξης Λισαβόνα που ζητάει κοινή πολιτική άμυνας και ε, συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά το ΟΑΣΕ η ύπατη εκπρόσωπο θα πρέπει να είναι παρατηρήτρια στον ΟΑΣΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, ε, οι πολυμερείς οργανισμοί είναι περίπλοκοι όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γίνονται όλες οι διαδικασίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές προσαρμογές έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης να μπορεί να κυρώνει και να κυρώσει συμφάσεις ε, προκειμένου την ΕΣΔΑ την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ε, ξέρουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ε, ιδιαίτερο στο χαρακτήρα του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα λέει και η συνθήκη αυτά. Και άλλος ε, πολυμερής οργανισμός, σας είπα, είναι ο ΩΣΑ και η Ευρώπη να μην είναι μόνο παρατηρητής, αλλά πλήρες μέλος. Και πάλι είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες και συντρέχουσες αρμοδιότητες που είναι στον όσα. Έκτον, και άλλο περίπλοκο θέμα και πιο ασταθές. Είναι η διπλωματία των συνόδων κορυφής, το G20 και το G8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κανονικά να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες και πλήρως να εκπροσωπείται αλλού σε συνεδριάσεις ε, του G7 των Υπουργών Οικονομίας. Και το G20 επίσης ε, κερδίζει όλο και περισσότερο σε σημασία και σε επιρροή. Γι' αυτό θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε υπουργικό επίπεδο στις υπουργικές ε, συνόδους κορυφής του G20. Αυτά είναι τα έξι κεφάλαια που σας είπα, έξι ενότητες τις οποίες επικεντρώνεται το σχέδιο εκθεσής μου που βεβαίως ε, είναι στη διάθεσή σας και για τροπολογίες και για τις δικές μου τροπολογίες και απομένουν πολλά στοιχεία να διευκρινιστούν, να συγκεκριμενοποιηθούν, να δοθούν νέες ιδέες. Θέλω να ευχαριστήσω, όπως περιπτώσει, το Ίδρυμα Αλτερνατίβα εναλλακτικέ για τη μελέτη που εκπώνησε και νομίζω ότι σας έχει διανεμηθεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρή έκθεση, πάρα πολύ αντικειμενική και αυστηρή με ε, νέες ιδέες χρήσιμες για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να λάβει θέση σε αυτό το περίπλοκο θέμα που για πρώτη φορά μας απασχολεί και σε μια στιγμή που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Πίτερ Βάσκετ και τον, ε, τη γραμματεία της έκθεσής μας για τη συστηματικοποίηση και για τις συνέργειες που έφερε σε αυτή την έκθεση πολιτικά ασχολούμαι με αυτό το θέμα και από τη γραμματεία για τη ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα προσπαθήσω ο συντονισμό που καμιά φορά λείπει μεταξύ κρατών μελών και θεσμικών οργάνων να επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μα μεταξύ των διαφόρων ε, ε, στοιχείων που μας απασχολούν ενός με τους διάφορους πυλώνες. Θα ήθελα να απευθυνθώ και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολούνται με αυτά τα θέματα τη πολυμερούς συνεργασία. μας βοήθησαν πάρα πολύ για να έχουμε μια συνολική θεώρηση ε, του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διάφορους οργανισμούς και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους βοηθούς μου και τους συνεργάτες μου που είχαν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους αλλά εργάστηκαν θαυμάσια για να μπορέσουμε να καταθέσουμε σχέδιο έκθεσης ε, πιο σύντομο από το αρχικό γιατί έχουμε τώρα κάποιες υποχρεώσεις, κάποιους περιορισμούς χρόνου και χώρου ε, για τη μετάφραση. Μας επιβάλλει ε, ορισμένο αριθμό χαρακτήρων σε μια ε, έκθεση η διοίκηση. Εγώ θα την ήθελα εκτενέστερη, τι να κάνουμε. Ελπίζω να τη βελτιώσουμε μέσω των τροπολογιών. Και με τους σκιώδεις ηγητές ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες, να κάνουμε την έκθεση αυτή είναι ενετική, διότι νομίζω ότι είναι θέμα θεσμικό. Αυτό που θα πρέπει να βγει από το Κοινοβούλιο είναι μια θέση του θεσμικού οργάνου. Και είναι σημαντικό και το περιεχόμενο και η ουσία και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια με παρουσία της κυρίας Άστον και στην ευρύτερη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή της στα διεθνή τεκτενόμενα. Είναι σημαντικό ε, η μεγάλη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική να γίνει ουσιαστική και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ε, διαδραματίζει το ρόλο που της αρμόζει και της αναλογεί διεθνώς. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Σα ευχαριστούμε κυρία Μουνής. Ε, θα δώσω το λόγο τώρα στους ομιλητές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Σας παρακαλώ να μην υπερβαίνετε τα δύο λεπτά κατά αγόρευση. Είναι πολύ φορτωμένη μέρη σε διάταξη. Η κυρία Χάουτα, από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θα χρειαστώ πάνω από δύο λεπτά. Κυρία Μούνη, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, μας παρουσιάσετε μια, ένα θαυμάσιο σχέδιο έκθεση και αυτό που λέτε να έρθει, είπατε, εκπρόσωπο οποίος ε, με μια, ένα λευκό έγγραφο για τις ε, πολυμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή τη στιγμή που εφαρμόζεται η συνθήκη της Λισαβόνας και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, έχει ορίσει τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία λοιπόν από αυτές πράγματι είναι να ενισχυθεί η πολυμέρεια. Αυτή είναι η στρατηγική ασφαλείας από το 2003. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της της ε, νομιμότητας με την ευρύτερη έννοια, να το συνδυάσουμε με τον εκδημοκρατισμό της παγκόσμιας διακυβέρνησης και πώς μπορεί να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την έννοια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό σχετίζεται άμεσα ε, με την έκθεση του ε, κυρίου Λάμπστορφ, την οποία και θα ακούσουμε σήμερα αργότερα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ε, συμμετοχή και έλεγχος των δραστηριοτήτων, ίσως με την ενίσχυση της Γενικής Συνέλευσης. Εξάλλου, όσον αφορά την νομιμότητα ε, της λήψης αποφάσεων ε, για την πολυμέρεια, ακούσαμε θαυμάσιες προτάσεις για το πώς οι νέε, ε, το G8 και το G9 μπορούν να εκπροσωπηθούν καλύτερα ε, στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ λοιπόν ε, βλέπουμε τον ενισχυμένο ρόλο των αδειόμενων δυνάμεων. Πράγματι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο, ισχυρότερο λέγιν στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ενισχύσουμε την περίφημη ερεσιμότητα και θα ήθελα να αναφέρω και το θέμα της εξορρόπησης των συμφερόντων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, αντισταθμίσουμε τα εμπορικά συμφέροντα με άλλα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και άλλα. Εδώ λοιπόν πρόσφατα το Κοινοβούλιο κατέθεσε μια θαυμάσια έκθεση που πρέπει να έχουμε κατά νου. Ε, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τους αναδυόμενους εμπορικούς μηχανισμούς ε, με πιο καινοτόμο τρόπο. Ας μην ξεχνάμε το Google αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σχετικά με το ότι η ε, λογοκρισία του διαδικτύου ε, στο, στην Κίνα μπορεί να αποτελεί και παραβίαση των διατάξεων του ΠΟΕ. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανοιχτή, με μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι το Συμβούλιο τη Ευρώπη, τη στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνεται να ε, συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν είχα κι άλλη να πω, νομίζω ότι τέλειωσε ο χρόνος μου. Σήμερα Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Λάμπστορφ τώρα, πρόεδρος ομάδας εργασίας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση της κυρίας Μουνής που τη βρίσκω πάρα πολύ καλή και θέλω να πω ότι εδώ πρόκειται για μια έκθεση η οποία κατά την άποψή μου ε, βασίζεται σε μια μελέτη την οποία έτσι ξεφύλει απλώς για να μιλικρινείς που κάνει όμως θαυμάσια εντύπωση. Ε, το θέμα τίθεται τελείως διαφορετικά ε, όπως πραγματικά ισχύει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Δηλαδή δεν μπορούμε να εμφανιστούμε με τον ίδιο τρόπο σε όλους αυτούς τους ε, διεθνείς οργανισμούς και αυτό αναφέρεται πάρα πολύ καλά στην έκθεση. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η καθυστερημένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά καθυστερημένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οργανισμούς είναι ένα πρόβλημα. Και στα αγγλικά πολλές φορές λέμε ε, πράγματι υπερεκπροσωπούμεθα αλλά υπολειτουργούμε. Όντως, ε, πολλές φορές Δυστυχώ, ε, επειδή θέλουμε να εμφανιστούμε παντού, αυτό που κάνουμε είναι απλά να περιζόμαστε σε δραστηριότητε συντονισμού. Και θέλω να πω τα εξή. Όσον αφορά την κατεύθυνση, πράγματι τη συμμερίζουμε. Πολύ καλή η ανάλυση στη μελέτη. Ε, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, ίσω να καταστήσουμε την έκθεση περισσότερο πολιτική. Γιατί όπω είπε και η κυρία Χάουταλα, έχει φτάσει πια η κατάλληλη χρονική στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή βέβαια μια κρίση, γι' αυτό και η συζήτηση αφορά περισσότερο ε, τους ε, αφεκιονάντους αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα. Όμως εδώ υπάρχει και ένα πολιτικό μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Άλμα πρέπει να κάνουμε, σαφέστεροι να είμαστε στα αιτήματά μας και προς τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, κυρίως όσον αφορά τον απολογισμό και την υποβολή συστάσεων. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει και από τη συνάντησή μας. Προτείνω πιο συγκεκριμένα τα εξή να διαγραφεί το εδάφιο Α, γιατί θεωρώ ότι το Β είναι πάρα πολύ καλό. Το Α μας δίνει έτσι μια ακαδημαϊκή ιδέα για τις διάφορες διαδικασίες ε, της ε, παγκοσμιοποίησης και τις συστημικές αποτυχίες αυτών των προσεγγίσεων. Εγώ θεωρώ ότι η παγκοσμιοποίηση είναι περισσότερο μια ακαδημαϊκή κουβέντα. Όμως το εδάφη ήταν μια θαυμάσια διατύπωση που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για ε, είσοδο στο θέμα, για προήμιο στο θέμα. Κατόπιν, δεν ξέρω κατά πόσο πράγματι έχει λάβει η χώρα η μεταρρύθμιση στην Παγκόσμια Τράπεζα στο Διεθνές Δομινικό Έχει λάβει χώρα αυτή η τροποποίηση ξέρω όμως για την Παγκόσμια Τράπεζα. Κατά τα άλλα, ίσως θα βοηθούσε να ε, επισημάνουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται θαυμάσια μέσα στην πολυμέρεια. Είναι η ε, επιχείρηση Αταλάντα όπου είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Αυτές ήταν οι πρώτες παρατηρήσεις. Θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά έχει σημασία η κατευθυντήρια, η κατεύθυνση που αναλαμβάνει που ακολουθεί, με συγχωρείτε, η έκθεση και αυτή κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε κύριο Σκούκεν τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι σύντομος. Το αντικείμενο της έκθεσης είναι τέτοιο ώστε δεν υπάρχουν αντικρούμενα σημεία. Όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Θέλουμε να έχει ηγετικό ρόλο η Ένωση. Δεδομένου των τραγικών εξελίξεων στη διεθνή πραγματικότητα που βιώνουμε σχάτως, είναι λογικό αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ε, σε, με ισότιμους όρους να μάλλον να έχει την ίδια θέση όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα, την ίδια θέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες δηλαδή εκ των έσω πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας και να αναβαθμίσουμε τη θέση μας σε διάφορους ε, διεθνούς ε, οργανισμούς. Η έκθεση της κυρίας Μούνης ε, είναι μια καλή βάση, ένα καλό έρισμα για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Συμφωνώ και με τους συναδέλφους από την Ισπανία. Δεν είναι ακαδημαϊκή η θέση τους, δεν είναι θεωρητική, αλλά τουλάχιστον κάνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις. Και αυτό είναι το γενικότερο μου σχόλιο για το ψήφισμα. Δηλαδή, έχουμε πάρα, πολύ, πάρα πολύ ωραίες ιδέες, ίσως και υπερβολικά πολλές ιδέες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα το έγγραφο, πρέπει να είναι ρεαλιστικό το σχέδιό μας. Να εκπονούμε μια πολύ ε, ουσιαστική πολιτική, να βρούμε τις λύσεις για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Δηλαδή τέτοιου είδους ψηφίσματα είναι τόσα, τόσο πολύ άριθμα αυτά τα ψηφίσματα και δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε απτά αποτελέσματα ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσω του ψηφίσματος. Σας ευχαριστούμε, κύριος Presidente. Eh, ehm, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Συγήτρια για την έκθεσή της. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ έτσι κάπως ε, γενικότερα, κυρίως ε, διότι πιστεύω ότι η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, έχει περισσότερο μια ε, προσέγγιση διακυβερνητική. Η αλήθεια είναι ότι η παγκοσμιοποίηση οδήγησε στο να χάσουμε σημαντικά στοιχεία της εδαφικής της κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Κυρίως αυτό αφορά στα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι βέβαια ότι ε, δεν ξέρουμε κατά πόσον ε, πράγματι πρέπει η εθνική κυριαρχία να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, να εκχωρηθεί ε, κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως κάποια στοιχεία αυτής χάνονται και ο μόνος τρόπος για να τα ανακτήσουμε είναι να την διαχειριζόμαστε με δική μας συγκατάθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούμε απλά και μόνο επειδή η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το σκληρό ε, και συμμετέχει κανείς σε αυτή την παγκοσμιοποίηση με μέσα και εργαλεία τα οποία συγκρίνονται με αυτά που διαθέτουν οι άλλες ε, μεγάλες χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό πρέπει κανείς να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ε, και να το λαμβάνει υπόψη του. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ο εκδημοκρατισμός εκδημοκρατισμός ε, των διεθνών οργανισμών ε, και αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Ε, όχι μόνο τον εκδημοκρατισμό, αλλά αν θέλετε και τον εξορθολογισμό. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όλοι οι θεσμοί του Bretton Woods, δηλαδή η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πρέπει να ενταχθούν στο ίδιο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και επίσης και, στον, και ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και αυτός πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα. Ε, γιατί θα πρέπει βεβαίως και να δίνονται κίνητρα αλλά και να επιβάλλονται και πρόστιμα, κυρώσεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα από το σύστημα, το διεθνές σύστημα. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Και με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει πράγματι να συμμετέχει περισσότερο στον εκδημοκρατισμό αλλά και στον εξορθολογισμό των διεθνών οργανισμών έτσι ώστε πράγματι να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκόμες τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Μαρία Μουνίσε για το εξαιρετικό ψήφισμα που μας υποβάλλει. είναι πλήρες, εντοπίζει τα προβλήματα και προτείνει λύσεις. Η Μαρία προσπάθησε να προτείνει μετριοπαθείς λύσεις ώστε να συλλέξει και τη συνένεση των μελών. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας, ε, ή μάλλον να θέσω αλλιώς. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο θάρρος ε, στο Κοινοβούλιο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα και για να προτείνουμε ε, αποτελεσματικές λύσεις εξηδίας εμπειρίας. Ε, θα έλεγα ότι η μεταρρύθμιση του κογουαστορικού κανονισμού του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει κέρια σημασία. Τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις προβλέψεις και τους στόχους που συνεπάγεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά. Αν είμαστε πιο θαραλοί, αν πιέσουμε για την τροποποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την διαδικασία, αν συμφωνήσουμε μεταξύ ημών, για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπούμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα Δεν πρόκειται για μια επανάληψη των θέσεων μα ένα διευρυμένο δηλαδή συμβούλιο να έχει έδρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έλεγε η Μαρία. Ναι, σημαντικό και αυτό, αλλά είναι ο ελάχιστος κοινό παρονομαστής. Ε, περισσότερα θα έπρεπε να επιδιώκουμε. Αν δεν έχουμε εμεί το όραμα, αν δεν αναλάβουμε εμεί ηγετικό ρόλο στο Κοινοβούλιο εννοώ, ποτέ δεν πρόκειται να προκύψει αυτό από τα κράτη-μέλη. Γιατί βρίσκονται και σε απόγνωση τώρα, πώς να το πω αλλιώς. Πρέπει να είναι πιο θαραλέο το κοινοβούλιο, να συζητήσει τη διεύρυνση, τη δέουσα εκπροσώπηση, τι συνεπάγεται αυτός προ τις ευθύνε μας. Βρίσκω ότι είναι ενδιαφέρον και μάλλον ανησυχητικό που τρεις επιδιώκουν μόνιμη θέση, η Βραζιλία, η Ινδία και η Γερμανία και αυτές οι τρεις δυνάμεις απίσχαν από την ψηφοφορία στο ψήφισμα για την παρέμβαση στη Λιβύη. Δηλαδή, τι, θέλουν την ευθύνη, θέλουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο ασφαλεία και όταν υπάρχει κρίσιμη ψηφοφορία επιλέγουν την αποχή. Πρέπει να ε, είναι πιο καταλητικό, πιο αποφυστικό ο ρόλο μας. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε εμεί την αποχή. Για το ΒΕΤΟ, την αρνησή κυρία, δεν μπορεί να υπάρξει ε, πραγματική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας αν δεν αναθεωρηθούν ε, τα περιβέτο, γιατί ε, παραλύει το Συμβουλίο Ασφαλείας συχνά λόγω του βέτο. Υπάρχουν και άλλα πολύ εύστοχα στοιχεία μέσα στην έκθεση, αλλά θέλω να είμαστε πιο θαραλέοι, πιο τολμηροί στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα κάνω σχετικές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέλε. Äh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Μινής ε, για την έκθεση που μας ε, παρουσίασε. Εγώ θα ήθελα ε, να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο παραγράφους, καταρχήν στα σημεία υπερθυμών 11 και 12. Βεβαίως υποστηρίζω κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα το σημείο 11 ως έχει. Ελπίζω μόνο επιτόπου όσοι λάβουν τις αποφάσεις την επόμενη φορά να μεριμνήσουν καλύτερα. Δηλαδή, όταν θα τεθεί το θέμα του να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει το λόγο στη Γενική Συνέλευση, ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα οργανωμένα. Θέλω να ελπίζω ότι αντλήσαμε διδάγματα από τα λάθη μας ε, όταν ήμασταν στην Κινσάσα, στην συνέλευση των ΑΚΕ ε, η Υπουργό Ασκογιάννα εξήγησε ακριβώς ε, τι θα γίνει και αυτό ήταν απαράδεικτο. Δηλαδή, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία ημέρα πριν από την ψηφία στην Κογιάννα εμφανίστηκε εκεί και είπε αύριο ε, θα ψηφίσετε προφανώς ως ομάδα ΑΚΕ από κοινού με Αυτό έγινε μία μέρα νωρίτερα και είπανε μα με συγχωρείτε εμείς διαφορετικά ε, σχηματίζουμε άποψη. Δεν γίνεται από σήμερα σε αύριο να κάνουμε αυτό που θέλετε και τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ελπίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και ελπίζω στο μέλλον να υπάρχει και καλύτερη οργάνωση. Νομίζω λοιπόν ότι στο σημείο 12 θα πρέπει εκεί να είμαστε λίγο περισσότερο φιλόδοξοι. Και όχι μόνο να καλούμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εξηγούν στους άλλους τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, καλό και αυτό, όμως ε, πιστεύω ότι από τότε που έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και από τότε που θέλουμε ή αποφασίσαμε να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, οφείλουμε να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση που θα οδηγήσει στο τα κράτη-μέλη τα οποία εκπροσωπούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εκπροσωπούν την γνώμη όλων. Όπως ακριβώς κατορθώνουμε στο Συμβούλιο Υπουργών να επιτύχουμε κοινέ θέσει ή και σε άλλα συμβούλια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ε, θα πρέπει ε, να γίνεται και το ίδιο ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Να υπάρχει κοινή στάση στις ψηφοφορίες. Και εδώ πρέπει να σας πω, δεν έχω υπόψη μου μόνο αυτό που έκανε η κυβέρνησή μου στην ψηφορία για τη Λιβύη, το, το, θέτω το θέμα έτσι κάπως γενικότερα. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Μονίθ για την έκθεση αυτή, το σχέδιο έκθεσης που πραγματικά στόχο έχει να αναβαθμίσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς. Με κάλυψε ο κύριος Κούκαρ, εκπρόσωπος της ομάδας μου. Θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή αποτελεί καλή βάση για να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας. Θα ήθελα να κάνω όμως μερικά σχόλια εγώ σε σχέση με δύο οργανισμούς ασφαλείας. Ο ένας αυτός ο οργανισμός είναι το ΝΑΤΟ το Κοινοβούλιο παίζει εξέχοντα ρόλο στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και το άλλο έχει να κάνει με τη συνεργασία που έχουμε στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Προχθές είχε έρθει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ και συνεργαζόμαστε θαυμάσια για παρατηρήσεις εκλογών, τέτοιες αποστολές με ορισμένα προβλήματα, αλλά α, αυτά τα ατού που έχουμε και εμπειρία από τη συνεργασία θα πρέπει να τα λέμε και στην έκθεση. Και τέλος, κάτι που έχει να κάνει με τη συνεργασία στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε αρνητική ε, εμπειρία ε, που δεν κατάφερε να εκλεγεί Ευρωπαίος Πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση. Δεν ε, ανταποκρίνεται η κατάσταση στα νέα χαρακτηριστικά της Σύνθηκης Λισαβόνας. Νομίζω θα πρέπει να αποκομίσουμε αυτές τις εμπειρίες και αυτό που είπε ο κύριος Γκάλερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι πραγματικά αξιοθρύνητο το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ψηφίζουν προς την ίδια κατεύθυνση και δεν ευθυγραμμίζονται. Αυτό δεν θα ε, σήμαινε ένα ελάχιστο συντονισμό εκ των προτέρων στα τόσα λίγα μέλη που έχουμε εκεί. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούγεται με μία φωνή. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ επιθυμητό. Ε, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Λάμστορφ για την αιτιολογική σκέψη Α, γιατί είναι κάπως ανητική διατύπωση και το κεφάλαιο για τα Ηνωμένα Έθνη είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους της χιλιετίας και τη σημαντική χρηματοδοτική εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οργανισμό αυτό πρέπει να τονιστούν και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ισχύσουμε το καθεστώς μας. Τελειώνω, Πρόεδρε, είναι καλή βάση, επαναλαμβάνω, πηγαίνει σωστή κατεύθυνση και όπως είπε και η κυρία Μουνίθ, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονιζόμαστε και οι ίδιοι με τρόπο αποτελεσματικό. Έψαχνα ε, στα έγγραφά μου την ισπανική έκδοση της έκθεσης και τα βρήκα μόνο στα αγγλικά. Ξέρει η κυρία Μουγής ότι θα πρέπει να μοιράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες εκθέσεις αυτές. Ελπίζω να διορθωθεί αυτή η ανομαλία σύντομα. Euh, Ευχαριστώ. Σε όλες τις γλώσσες θα έχουμε την έκθεση την ώρα που θα ψηφίζουμε τις τροπολογίες. Μαθαίνω. Ο κύριος Γκυμαράες έχει το λόγο τώρα. Σύμβουλος για θέματα σχέσεων σε πολυμερείς οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο υπόψη. Θα μιλήσω λοιπόν για το, το σχέδιο της έκθεσης. Νομίζω πρέπει να συγχαρούμε ε, την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το θέμα και πράγματι ε, προσπαθεί ε, να εντάξει και το πνεύμα και το νόημα την ουσία της συνθήκης Λισαβόνας. Το γράμμα και το πνεύμα. Πράγματι λοιπόν ε, ε, το ψήφισμα αυτό ήταν πολύ δύσκολο να περάσει τη Γενική Συνέλευση και αν ε, λάβουμε υπόψη μας ε, το σχέδιο αυτό της έκθεσης ε, ήταν κάποιο δευτερεύον ε, θέμα το οποίο μπορεί βέβαια να λυθεί και αυτό είναι το δικό μου το καθήκον. Αυτή όμως η έκθεση δίνει μια γενική εικόνα της κατάστασης ε, και αυτό είναι πολύ καλό. Δείχνει ότι υπάρχει ένταση και δυσκολία από πλευράς κρατών μελών να ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση. Και υπάρχει επίσης και πίεση πίεση για την αναδιάρθρωση της ε, παγκόσμιας ε, διακυβέρνησης. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν το ρόλο τους στους πολυμερείς, στα πολυμερή φόρουμ είναι σαφές ε, ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό στην πρακτική. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα του Μοντής είναι της ε, νομικής οντότητας. Το γεγονός ότι είμαστε παρατηρητές σε πολυμερή φόρουμ, η φόρα είναι το σημείο εκκίνησης. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ευτής από την αρχή λοιπόν θελήσαμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερο ρόλο στους διεθνείς οργανισμούς και για μας η πρόκληση είναι πώς μπορούμε να επεμβαίνουμε στα πολυμερή φόρα. Αυτό το έθιξαν πολλοί ομιλητές και αναφέρεται και στο σχέδιο έκθεσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ε, πολύ υποβαθμισμένη θέση, τη θέση του παρατηρητή. Πιο συγκεκριμένα θέλω να πω ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να γίνει μια συζήτηση τον Ιούνιο. Εκεί θα συμμετάσχουμε ενεργά. Θα είναι ο ρόλος των ΗΕ στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλεία, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ε, δείγματα πρόοδου θα μπορούσαν να προκύψουν από το να εστιάσουμε την προσοχή μα στι ε, μεθόδου εργασία του Συμβουλίου Ασφαλεία. Αυτά είχα να πω. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριος ο πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση για τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, οπότε θα ασχοληθούμε με το κομμάτι τη έκθεση που αφορά σε αυτό το τομέα πολιτική. Ε, η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στη συζήτηση για τα οικονομικά στη διεθνή σκηνή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, είμαστε από τι μεγαλύτερε οικονομίε του κόσμου και το ευρώ είναι ένα από τα σημαντικότερα νομικά νομίσματα. Η ζώνη ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να έχουν ηγετικό ρόλο στις πολυμερείς οργανώσεις και στη διεθνή σκηνή. Η ενιαία φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακουστεί και γι' αυτό καλωσορίσουμε το ψήφισμα της κυρίας ε, Μιονής και τις συστάσεις της. Η τωρινή κατάσταση πόρο απέχει από το ικανοποιητικό επίπεδο όπως ανέφερε και η συγγετρία και οι εμπειρογνώμονες. Είναι μάλλον πολιτικό το ζήτημα και γι' αυτό καλωσορίζουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία παρατηρήσει θα κάνω. Έχουμε το άρθρο 138 της συνθήκης που προβλέπει την ακολουθητέα διαδικασία ώστε να εξασφαλίσουμε εκπροσώπηση τη ζώνη ευρώ στους διεθνεί χρηματοπιστωτικού οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά πρέπει να προτείνει την συγκρότηση της εκπροσώπης που θα εγκρίνει μετά το Συμβούλιο αυτή τη διαδικασία. Στις 20 Οκτωβρίου 2010, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 225 της Συνθήκης, ε, αναφέρεται το δικαίωμα πρωτο, πρωτοβουλίας ε, και άρα μας ζητήθηκε βάσει του άρθρου 138 να καταθέσουμε πρόταση πρωτοβουλίας ώστε να ενισχύσουμε την εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ. το ψήφισμα της κυρίας Μιονής νομίζω θα μπορούσε να παραπέμπει σε αυτό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου γιατί από αυτό προκύπτει και η νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Εν συντομία, ε, μήπως ήθελαν οι εμπειρογνώμονες το λόγο για να σχολιάσουν την έκθεση. No. No. τότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τα επικοδομητικά του σχόλια για το σχέδιο έκθεσής μου. Όλοι βεβαίως από τις διαφορετικές πολιτικές σκοπιές αλλά και από τη θεσμική σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα φροντίσουμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε το σχέδιο έκθεσης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πρόβλημα χώρου, ουσιαστικό, περιορισμούς. Γι' αυτό περιορίστηκα εγώ στο να κάνω προτάσεις παρά να ε, επαναλαμβάνω αυτά που ήδη συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Αν και τα είπαμε η συνεργασία του Κοινοβουλίου με διάφορα άλλα θεσμικά όργανα, ε, ε, τι δεν γίνεται καλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αξιοποιούμε τον περιορισμένο χώρο που έχουμε για να κάνουμε νέες προτάσεις και να επισημαίνουμε τι πρέπει να λυθεί. Επίσης, συμφωνώ ότι η αιτιολογική σκέψη α μπορεί να είναι λίγο απότομη στη διατύπωσή της για την παγκοσμιοποίηση και μπορεί κάπως να απαλληλθεί με κάποιες αποχρώσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση συντάχθηκε στα αγγλικά αρχικά γιατί λόγω των προθεσμιών για να μπορέσουμε να φτάσει στην Ολομέλεια που θα συζητηθεί και παρουσία της κυρίας Άστον όταν θα εγκριθεί και η έκθεση Αλμπερτίνη για την εξωτερική πολιτική δεν προλαβαίναμε να τη γράψουμε σε άλλη γλώσσα για να μεταφραστεί Γι' αυτό δεν την έγραψα στα ισπανικά, την έγραψα κατευθείαν στα αγγλικά για να έχουμε ένα πρώτο σχέδιο, κατανοητό υποθέτω, ελπίζω από όλους ε, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες εκδόσεις σε όλες τις γλώσσες μας και βεβαίως και στα ισπανικά. Και οι τροπολογίες προφανώς θα έρθουν σε όλες τις γλώσσες. Είναι λοιπόν ένα πρώτο σχέδιο έκθεση και επειδή μα πίεζαν οι προθεσμίε και είχαμε καθυστερήσει στη σύνταξη, γι' αυτό άλλωστε το λόγο είναι και στα αγγλικά. Επαναλαμβάνω για να μπορέσουν να την καταλάβουν όλοι πριν φτάσουν οι μεταφράσεις. Για τα υπόλοιπα σχόλια νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει αυτό καλή βάση για συνένεση στην Επιτροπή μας και η έκθεση τελικά να είναι όσο γίνεται πιο προσανατολισμένη και ευθυγραμμισμένη με τις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες, τα όνειρα, τα οράματα της Επιτροπής μας για την εξωτερική πολιτική και τα όσα ορίζει η ε, συνθήκη της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή στους διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σαλαφράνκα, ζητήσατε πάλι το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να, να αναφερθώ στο γλωσσικό. Εμείς δεν είπαμε να μην συζητηθεί σήμερα επειδή δεν είναι μεταφρασμένη έκθεση. Αλλά αυτό δεν είναι στη διακριτική ευχαίρεια του εισηγητή ε, ότι μας κάνει και χάρη, ε, το γράφει σε μία γλώσσα και μετά θα το φέρει και σε άλλη γλώσσα, ας πούμε, το κείμενο. Δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία. Το είδαμε και στο θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Οι κανόνε θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις ε, εκδοχές, τι γλωσσικές εκδόσεις να τις έχουμε, είτε είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, δεύτερη, τρίτη, τελευταία. Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο αποφασίζει ο εισηγητή. Δεν θελήσαμε να ε, ε, βάλουμε εμπόδια στη συζήτηση, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, αλλά δεν είναι δικαιολογία ότι πιέζουν οι προθεσμίες. Οι προθεσμίες είναι γνωστές για όλους, είχαμε πολλές ευκαιρίες και θα ε, έπρεπε να έχουμε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις. Εντάξει, τώρα θα δουλέψουμε το αγγλικό κείμενο, αλλά θέλω να το πω για να ακουστεί κάποια στιγμή να ε, εφαρμόζουμε τους κανόνες όπως αυτοί ισχύουν. Ευχαριστώ. Μου είπαν ότι το σχέδιο ψηφίσματος θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών. Το χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, για την υποβολή των τροπολογιών ε, Μαρτίου στις 12, δεύτερη συζήτηση στην Επιτροπή μας στις 19 Απριλίου, ψηφοφορία στις 20 και το Μάιο θα περάσει από την Ολομέλεια. Θα συζητηθεί στην Ολομέλεια το θέμα. Μετά, περνούμε στο επόμενο σημείο και θα καλωσορίσουμε την κυρία Φραντσέσκα Μπαλτσάνη που φέτος είναι η συγγήτρια για τον προϋπολογισμό 2012, για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού 2012. Ε, να συναντηθεί με τους εκπροσώπους όλων των καθήλια αρμοδίων επιτροπών, ώστε να λάβει υπόψη τα συγκεκριμένα σχόλιά τους όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού και κατόπιν συζητηθεί προς έγκριση από ε, τις συναρμόδιες ε, δημοσιονομικές αρχές, δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι σχετικά με τη δυνατότητα η Επιτροπή Προϋπολογισμών να εγκρίνει τις προτάσεις της δικής μας Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τον Προϋπολογισμό το 2012. Είμαι επίσης πεπισμένος πως η κυρία Μούνης που είναι αρμόδια για τη σύνταξη της έκθεσης, της νομοδότησης μάλλον για την έκθεση της κυρίας Μπαλτσάνη, με την ιδιότητα της σκιώδουση της θα μπορέσει να υπεραμεινθεί των καταλληλότερων προτάσεων δοθήσεις και της διεθνούς συγκυρίας, διότι χρειάζονται επιπρόσθετη πόροι σε διαρκή βιώσιμη βάση. κυρία Μπαλτσάνη. Grazie Presidente. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για αυτή τη συνάντηση. Πέρυσι λοιπόν ε, κάναμε την εξής εμπειρία. Η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, παρότι τυπικά υποτίθεται ότι απλούστευσε τη διαδικασία του ε, προεπολισμού, γιατί περιόρισε κατά μία τις συνδιαλλαγές, παρόλα αυτά κατέδειξε ότι ο προϋπολογισμός πάντα συνοδεύεται με πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά λεπτά θέματα. Εφέτος λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό ευθύς εξ αρχής να διαβουλευτούμε με τις επιτροπές έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι το θέμα του προπολογισμού δεν θα παραμείνει μόνο στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά θα επηρεαστεί το θέμα και από τις ε, συνεισφορές των υπόλοιπων επιτροπών. Φέτος λοιπόν η δική μου η πρόταση είναι να συμπεριλάβουμε τις προτεραιότητες για το 2012 στην στρατηγική του 2020. Ε, το στο πλαίσιο λοιπόν της στρατηγικής 2020, γιατί δεν πρόκειται μόνο για μια πολιτική επιλογή επενδύσεων σε ε, μέσο μακροπρόθεσμο ε, πλαίσιο, αλλά και διότι μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ε, πραγματικά ευρωπαϊκές προτεραιότητες, προτεραιότητες που είναι ουσιαστικές και προτεραιότητες τις οποίες συμμεριζόνται και τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν αυτό το θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τα κράτη-μέλη καλούνται ε, να συμμετάσχουν ε, σε αυτή τη στρατηγική. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και εντάσσονται διαβουλεύσεις ε, με τις ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε με βασιστικές αρμοδιότητες ποια είναι τα πιο λειτουργικά στοιχεία που ε, θα συμβάλλουν στην επίτευξη και χάραξη της στρατηγικής 2020. Αυτή λοιπόν η Ειδική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα για πάρα πολλά πολιτή ε, προγράμματα ε, ορισμένα, σε ορισμένα εξ αυτών υπήρξε, υπήρξαν θετικής, θετικές εξελίξεις έχουμε κυρίως, έχω κυρίως κατά νου την πολιτική γειτονίας όπου αυξήθηκε κατά 10% η χρηματοδότηση χρηματοδότηση ε, σε σχέση με την αρχική. Υπήρχαν όμως και αρνητικές εξελίξεις ε, ε, προγράμματα που περικόπηκαν κατά πάνω από 20%. Πάντως αυτή η Επιτροπή είναι αρμόδια και για τα κονδύλια του Ταμείου Έκτακτων ε, Συνθηκών. Εκεί υπάρχει κάποια ευελιξία στον προπολογισμό μας, μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου έχει ευελιξία. Έτσι λοιπόν αυτή εδώ η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στο να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε, την ευελιξία. Αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να διευκρινίσουμε τις ε, προτεραιότητες που μπορεί να προτείνει η Επιτροπή αυτή για την κατάρτιση του προπολογισμού. Και θέλω να πω ότι οι ίδιες αυτές προτεραιότητες θα μας οδηγήσουν στο να ορίσουμε και τα προγράμματα πιλότους ε, κατά την ε, προετοιμασία. 3 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να έχουμε έστω ένα προσωρινό κατάλογο ε, των προγραμμάτων αυτών και να υπάρξει και μία πρώτη αντίδραση. Πάντως θα είναι και η ίδιες προτεραιότητες οι οποίες με διαφανή τρόπο μπορούν να μας οδηγήσουν στο να ορίσουμε τις τροπολογίες εκείνες ε, που θα το κάνουμε όταν θα κληθούμε να ορίσουμε ε, συγκεκριμένα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, όσον αφορά στον προπολογισμό. Έτσι λοιπόν, σας καλώ το θέμα του προπολογισμού να το εντάξετε στο επίκεντρο των συζητήσεών σας για να διασφαλιστεί ότι πράγματι θα έχουμε κοινή στάση στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διασφαλιστεί επίσης ε, ότι από εκεί θα καθορίσουμε και εμείς ε, τη στάση μας για το σχέδιο ε, προϋπολογισμού ε, μέχρι τις 20 Απριλίου. Οι τροπολογίες πρέπει να είναι σαφείς, διαβανείς και πρέπει να συμβάλλουν με τρόπο αποτελεσματικό και χρήσιμο. Έτσι λοιπόν η μπάλα αν θέλετε περνάει στη δική σας την Επιτροπή και θέλω να πιστεύω ότι θα λάβετε υπόψη στο θέμα το δικό μου, το θέμα του προπολογισμού, με τη δέουσα προσοχή. Η κυρία Μουνής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έκθεση ε, του προπολογισμού είναι ακόμα πάρα πολύ πρόωρο για να κάνουμε εξαντλητική ανάλυση. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια κυρία Μπαλτσάνη ότι η εστίαση θα πρέπει να συνδέεται με τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας που είναι η ανεργία και η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική του 2020. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε ε, τις ε, προοπτικές για τη χρόνια υποχρηματοδότηση από την οποία πάσχει η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε παγκόσμιος πρωταγωνιστής και έχουμε ευθύνη να χρηματοδοτούμε ε, τις διεθνής ε, δράσης μας ε, και υπάρχει κίνδυνος να περιοθεροποιηθούμε εάν δεν είναι σωστή η παρουσία μας. και αν υποχρηματοδοτείται χρόνια η πολιτική μας κάτω των αναγκών της, η Ευρώπη αυξάνει σημασία σήμερα και δεν νοείται προϋπολογισμός που να μην ε, συνάδει με αυτά τα δεδομένα. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ακόμα τα ποσά και τα αριθμητικά στοιχεία θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο να αποφανθούμε σε λεπτομέρειες θα πρέπει να λάβουμε κάποια στοιχεία υπόψη μας, ωστόσο για τον προπολογισμό του 2012. Να σας πω τα διάφορα θέματα που θα πρέπει να ε, συμπεριληφθούν από τη σκοπιά της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει μια λύση στο πρόβλημα για το μέσο συνεργασίας με τις ε, ε, βιομηχανικές χώρες συν, δεν έχει νομική βάση πρέπει να δοθεί μια νομική βάση και σωστή χρηματοδότηση για στρατηγικούς τομείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Λατινική Αμερική. Μέγα τμήμα των χωρών αυτών της Λατινικής Αμερικής είναι κράτη με μεγάλη ανάπτυξη, με ε, αρκετή νομική ε, ασφάλεια στην ένωμη τάξη τους και θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το μέσο η ε, ICI-SIN. Επίσης, μας ανησυχεί η περικοπή που γίνεται στο μέσο σταθερότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιους καιρούς και αν υποπρικοδοτηθεί δεν θα μπορέσει να φτάσει στους στόχους του. Έχουμε επίγνωση των ε, δημοσιονομικών δυσκολιών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει ακριβώς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αυστηροί στις αναλύσεις και των διαφόρων ε, τίτλων του προπολογισμού. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας ε, στα εξωτερικά θέματα στη Μεσόγειο, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε στα όσα συμφωνούμε. Ε, αναθεωρείται πολιτική γειτονίας προς Νότον αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή θα πρέπει να είναι κίνητρο για να ενισχυθεί η πολιτική γειτονία προς τον Νότο με μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη ελαστικότητα και νέους μηχανισμούς στιβαρούς, κρατεούς και ε, βιώσιμους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία στην περιοχή. Γι' αυτό χαιρόμαστε για αυτά που λέει η Φραντσέσκα Μπαρτσάνη για το σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υποστήριξη των χωρών της Μεσογείου για να βοηθήσει στην οικονομική ε, δημοκρατική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως ορίζει παράγραφος 12 για τις κατευθείαν γραμμές της εισηγήτριας. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει για τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, τη δημοκρατία στη Μεσόγειο, να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, ευελιξία και στην Επιτροπή Εξωτερικών, να γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλες θέσεις του προπολογισμού, όχι ε, στον τίτλο 4, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή με ικανοποίηση σημειώνουμε ε, την ανακοίνωση 208 ης Μαρτίου ε, όπου ε, αναφέρεται μεγαλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια ως άμεση απόκριση, ενίσχυση του Frontex και ενίσχυση του εκδημοκρατισμού. Όλοι αυτοί οι στόχοι δεν θα πρέπει να παραμείνουν στα λόγια ε, αλλά να υλοποιηθούν στην ε, πράξη και προκειμένου στον προπολογισμό του 2012. Συμφωνώ επίσης με την εισηγήτρια ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εφαρμογή, καλύτερη εκτέλεση του προπολογισμού και επίσης να θυμίσουμε ότι στα τμήματα που αφαιρώνονται στην εξωτερική δράση, στον τίτλο 4, είναι πολύ υψηλή η απορρόφηση. Οπότε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το λύσουμε για το σύνολο του προπολογισμού, γνωρίζοντα όμω ότι αν πρέπει να μειωθούν κάπου κονδύλια, ε, αυτά δεν θα είναι εκεί που είναι ε, το maximum ε, η απορρόφηση και αυτή είναι εξωτερική πολιτική. Το ίδιο με τη στρατηγική 2020, για το 2020 αυτή μπορεί να είναι αξιόπιστη και σωστή μόνο εφόσον συνοδεύεται από την απαραίτητη χρηματοδότηση. Γιατί θα ήταν μεγάλα τα ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, χωρίς να επιβαρύνει ουσιαστικά τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στην έκθεση Φερνάντες στο διοικητικό τμήμα για τις δαπάνες των διαφόρων θεσμικών οργάνων έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες για να ε, δούμε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι επιπτώσεις θα έχει η λειτουργία ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης το 2012. Τα κράτη-μέλη κάνουν οικονομίες, αλλά χρειάζονται χρήματα για να τεθεί σε λειτουργία αυτή η υπηρεσία εξωτερική δράσης, για να είναι πραγματικά αποτελεσματική στη λειτουργία τη. Και ένα τελευταίο. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τις κατάλληλες δράσεις έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλύτερη και μεγαλύτερη προβολή προς τα έξω και να είναι ορατή. Δηλαδή τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγαίνουν σε άλλες οργανώσεις ή στα Ηνωμένα Έθνη σε διάφορα προγράμματα, έργα, σχέδια, οργανισμούς του ΟΗΕ θα πρέπει να τα προβάλλουμε, να γνωρίζουμε αν αυτό μπορεί να αθρηστεί στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θεματικές ενότητες ή απλώς αν είναι ε, υποχρεωτικές διεθνείς ε, χρηματοδοτήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει εκεί συνέργεια όμως και οι οργανισμοί αυτοί ε, να γνωρίζουν και να φαίνονται τα κονδύλια ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προβάλλεται καλύτερα και στο εξωτερικό. Όπως σας είπα, μέχρι να δούμε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα ποσά. Συζητάμε λίγο στον αέρα. Είναι πάρα πολύ πρόημο ακόμα το στάδιο για να κάνουμε πρόταση. Ε, ε, ε, αλλά ε, οι προσανατολισμοί είναι ακριβώς αυτοί που χρειάζονται και το είπαμε και στους κοιόδες εισηγητές, ε, γιατί είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους και με την εισηγήτρια της Επιτροπής Προεπολογισμών, στην οποία επίσης διαβίβασα τη θέση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμστορφ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Αφενό, ε, θέλω να σα ε, ευχαριστήσω που έρχεστε τόσο έγκαιρα στην Επιτροπή μα για να μάθετε ποιε είναι οι προτεραιότητε αυτή. Ελπίζω να κατάλαβα καλά ότι η συγγήτρια για τον προπολογισμό του 2012 ε, ασχολείται μόνο με τα εργαλεία του κοινωνικού προπολογισμού ο προϋπολογισμός του, ε, του ΕΡΔ συμπεριλαμβάνεται, ναι ή όχι. Με σχόλια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης του ΕΡΔ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ε, το εξής. Η παράκληση δική μου είναι και αυτό το ανέφερε και στην άρθρο κυρία Μουνής, ότι έχουμε ένα εργαλείο, ένα μέσο για την ε, προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω λοιπόν ότι το στοιχείο της προαγωγής της δημοκρατίας θα πρέπει να το προβάλλουμε έλαβε χώρα μια πολύ σημαντική συνάντηση με τους Αμερικανούς και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι μια σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάρα πολλές αρμοδιότητες, επίσης έχουμε μεγάλη αξιοπιστία διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα, όμως υπάρχουν και συνεχώς νέες προκλήσεις τις οποίες βλέπουμε να εμφανίζονται στη Βόρειο Αφρική. Εάν λοιπόν αυτή είναι η προτεραιότητα τότε ε, πράγματι θα πρέπει να την προβάλλουμε περισσότερο. Και εδώ αναφέρομαι και στην κυρία Μουνής. Ε, πράγματι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά αυτό το μέσο. Merci, madame. Ε. Ευχαριστώ, η κυρία Γιατεμάκη. Kiitoksia, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόλις τώρα λοιπόν ακούσαμε ε, διάφορες απόψεις τεκμηριωμένες και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη δική μου ε, την άποψη σε ορισμένα θέματα, κυρίως εκεί που διαφωνώ. Όσον αφορά στην πολιτική γειτονία. Η πολιτική γειτονία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι ε, του εξωτερικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, οι νότιες χώρες ε, να λάβουν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως ε, τώρα, όπου ελπίζω αυτό που γίνεται να είναι μετάβαση προς τη δημοκρατία. Παράλληλα, αυτή η οικονομική υποστήριξη προς την κατεύθυνση του Νότου δεν επιθυμούμε βέβαια να αφαιρέσει την υποστήριξη από τις χώρες που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι χρηματοδοτήσαμε κατά πολύ ε, τις ε, χώρες ε, του Μπενάλη και του Μουμπάρακ. Η Βόρειο Αφρική στηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως τώρα θα πρέπει τα κονδύλια να τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικότερα, να στηρίζουμε ε, τον εκδημοκρατισμό της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών, τα κονδύλια να δαπανώνται περισσότερο σε επίπεδο βάσης. Μέχρι τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πω ότι δεν τα κατάφερε και πάρα πολύ καλά. Το μέσο για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλύτερα για την υποστήριξη ε, της κοινωνίας των πολιτών ε, και στις ανατολικές και στις νότιες χώρες, αλλά και σε άλλα μέρη. Πρέπει να σας πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω ε, τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στον προπολογισμό από αυτήν την νέα πολιτική εκδημοκρατισμού. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν τις ε, ε, προεκτάσεις αυτής της νέας πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό είναι τελείως καινούριο για πολλούς από εμάς και το θέμα που τίθεται είναι πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί, ποια θα είναι τα επιπρόσθετα κονδύλια που θα χρειαστούν. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η περίφημη αιρεσιμότητα των κονδυλίων Partnership for Democracy and this Prosperity for Democracy, eh, Value for Money. Αυτά τα προγράμματα δηλαδή ε, τα οποία θα χρηματοδοτούνται εφόσον ε, πράγματι ενισχύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο εκδημοκρατισμός. Οι προτεραιότητες ε, του προπολογισμού είναι διαφορετικές από αυτές που μας απασχολούν εμάς. Παρ' όλα αυτά όμως και οι εξωτερικές σχέσεις θα πρέπει να ε, προβληθούν περισσότερο, να χρηματοδοτούνται καλύτερα. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική. Η Λατινική Αμερική υποτίθεται ότι θα είναι προτεραιότητα την ε, επόμενη χρονιά ε, και θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για τη Λατινική Αμερική. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να μετατοπιστεί λιγάκι το βάρος. Ευχαριστούμε κύριο Σφέρμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα απειχώντας κάποια σχόλια της κυρίας Μουνιές θα ήθελα να σχολιάσω τη Νότιο Μεσόγειο. Συναντηθήκαμε με την ομάδα παρακολούθησης ε, με τον κύριο Σαλαφράγκα την περασμένη εβδομάδα και μας απασχόλησαν τα οικονομικά εργαλεία. Πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, λόγω της νέας κατάστασης. Είναι σημαντικό για το 2012 να εστιάσουμε την προσοχή μας στο συντονισμό αυτών των εργαλείων. Πέρα από το πρόγραμμα γειτονία που υπάρχει, Συνεχίζεται και η διαδικασία για τη νέα εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που πρέπει να διευρυνθεί σε αυτή την περιοχή. Επίση, ε, συζητούμε για το EPRD και συνεχίζονται και συζητήσεις για διάφορα άλλα οικονομικά εργαλεία για την υγειοργική συνεργασία, για την επιστημιστική ασφάλεια, για την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να συντονίσουμε όλα αυτά τα εργαλεία για να μην υπάρξει επικάλυψη, να ενσαφίζει οι προτεραιότητες μας στη Νότια Μεσόγειο και για το 2012 και πιο μακρόπνοα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στην αιρεσιμότητα, να βρούμε τη σωστή μέθοδο που θα ακολουθήσουμε και για τα δημοκρατικά ζητήματα αλλά και για την διαχείριση των εργαλείων στήριξης για τη σωστή διαχείρισή τους. Επίσης πρέπει να αντεπεξέλθουμε στον εξής κίνδυνο. Υπάρχει τα, η αναλογία 2 3 1 τρίτο ανάμεσα στο βορρά και στο νότο της Ένωσης και αυτή η ισορροπία θα πρέπει να τροποποιηθεί αλλά με διπλωματικό τρόπο τόσο ώστε να βρούμε μια διέξοδο αποδεκτή για όλους. Κύριε Λάμστορφ, ε, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ασχοληθεί η κυρία Μπαλιτσάνη με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο αλλά υπάρχει η, μόνιμη, η προσωρινή επιτροπή Σουρή για τις δημοσιονομικές προοπτικές όπου θα ασχοληθούμε με αυτό και με άλλα ε, βασικά ζητήματα. Οπότε προτείνουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να παρακολουθεί τι εξελίξει τη ΣΟΥΡΕ. Ε, η 31η Μαρτίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στη ΣΟΥΡΕ πλησιάζει ο καιρό, και μετά θα συζητηθεί η έκθεσή μας για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο ενδιαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ήθελα μόνο να σας θυμίσω να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και στην ΣΟΥΡΕ. Σας ευχαριστούμε. Μία διευκρίνηση σε σχέση με την ερώτηση που έκανε η κυρία Γετεμάκη θέλω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το δημοσιονομικό αντίκτυπο της νέας εταιρικής σχέσης με τους ε, νότιους γειτονές μας. Ε, θα διαβιβάσουμε την ερώτηση, αλλά ε, δεδομένων των αλλαγών που έγιναν την τελευταία στιγμή στη μέση διάταξή μας, δεν εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα διαβάσουμε το ερώτημα. Κύριο Αλεφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω η Γενική Συγκίτρια για τον Προπολογισμό για την παρουσία Η κυρία Μονίθ έχει παρουσιάσει τις θέσεις δική μας επιτροπής. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ο κύριος Φάρμ τόνισε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες της νότιας όχθης Μεσογείου με τον επαναπροσανατολισμό τώρα της πολιτικής γειτονίας. Με ένα ζήτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή και θίγει πάρα πολλές ευαισθησίες στο θέμα της ε, νέας πολιτικής γειτονίας και παραπροσανατολισμού και ε, διοχέτευση των κονδυλίων από την πολιτική γειτονίας προς Ανατολάς και να τα στράψουμε προς τον Νότο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει και μια βαθιά αίσθηση ευελιξίας σε αυτά τα θέματα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό η ύπατη εκπρόσωπος να προσπαθήσει να συνδυάσει τα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο τα δημοσιονομικά που αφορούν σήμερα τη συζήτησή μας, αλλά και τα εμπορικά, τα οποία δεν θέτουμε στις εκχωρήσεις, παραχωρήσεις που σκεφτόμαστε αυτό τον καιρό, την αύξηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έναν προσανατολισμό των ε, ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά υπάρχουν ήδη όλα τα στοιχεία ε, και ε, οι προηγούμενες συμφωνίες πρέπει να τηρηθούν προς όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες. Και όπως λέμε σε μια ισπανική παροιμία, το θέμα δεν είναι να γδίσουμε ένα Άγιο για να ντύσουμε έναν άλλον, να τα πάρουμε από τον ένα να τα δώσουμε στον άλλον. Ε, αλλά ε, να αντιμετωπίσουμε τις επίγουσες ανάγκες που έχουμε στην άμεση γειτονία μας. Συμφωνώ με την κυρία... Ε, μάλλον Διαφωνώ πάρα πολύ με την κυρία Γιατεμάκη. Στη Λατινική Αμερική έχουμε πολύ μεγάλη παρουσία και στην Καραϊβική με συνόδους κορυφής αναπτύσσουμε και επεξεργαζόμαστε το αποτελέσμα της Συνόδου Κορυφής πέρυσι στη Μαδρίτη, θα πρέπει βεβαίως να σεβόμαστε και εκεί ε, τις ε, συμφωνίες μας και τις υποχρεώσεις μας. Στο μέλλον θα πρέπει να το σκεφτούμε σε βάθος. Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς, αλλά και από ποια χρήματα θα πρέπει όλα αυτά να συνοδεύονται. Στη συζήτηση πάντα για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Και να κάνω και μία σύσταση, Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να στρέφουμε όλα τα χρήματά μας προς τη νότια όχθη της Μεσογείου χωρίς να ξέρουμε τον προσανατολισμό τους. Γυρίσαμε μερικοί μόλις από την Αίγυπτο, στις 19 του μηνός έγινε ένα δημοψήφισμα και η αναθεώρηση του συντάγματος είναι στη γραμμή που ζητάει η μουσουλμανική αδελφότητα και το κόμμα του κυρίου Βάρα. Προσοχή λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε ε, παρόντε εκεί να βοηθήσουμε την κατεπίγουσα κατάσταση, την ανθρωπιστική βοήθεια, να πούμε ότι είμαστε διατεθειμένοι και στο μέλλον να βοηθήσουμε, χωρί να δεσμεύσουμε όμω του πόρου τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου, μέχρι να δούμε ποια κατεύθυνση παίρνει αυτή η υπόθεση. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ε, είμαι βέβαιο ότι η Υπηρεσία εξωτερική Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζονται, αλλά προσοχή πριν δεσμεύσουμε τα κονδύλια να ξέρουμε πού τα δίνουμε και ε, αν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ο δημοκρατισμός ή μήπως εκτροχιάζεται προς άλλες εναλλακτικέ ε, προτάσεις που δεν είναι ούτε δημοκρατικές ούτε σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών των χωρών αυτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαλζάνη, θέλετε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα από τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση και η πρώτη εντύπωση που αποκόμισα έχοντας ακούσει όλες αυτές τις ε, παρεμβάσεις είναι ότι όσον αφορά τον ε, τομέα 4 παρότι ίσως και να μην είναι ο σημαντικότερος τομέας του προπολογισμού, εκεί ε, εμφανίζονται περισσότερο τα προβλήματα που βέβαια μετά διοχετεύονται σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχουν ε, τα κονδύλια και να συνδυάζονται και με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εξάλλου, είναι απαραίτητο ε, να υπάρχει ευελιξία για να αναζητώνται και οι αποτελεσματικές απαντήσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Είναι επίσης απαραίτητο συντονισμού των μέσων ένας συντονισμός που είναι καθοριστική σημασίας όχι μόνο για να υπάρχει αποτελεσματικότητα τη στιγμή που τα κονδύλια γίνονται όλο και λιγότερο αλλά και για να υπάρχει συνέπεια και συνεκτικότητα στην υπεραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή εδώ όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτόν τον τομέα που αναμφίβολα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα υποχρηματοδότησης. Και σίγουρα από αυτόν τον τομέα θα κληθούμε να απαντήσουμε σε θέματα που έχουν αλλάξει, όπως το θέμα της Μεσογείου. Η παρέμβαση στη Μεσόγειο είναι ένα θέμα ε, που επηρεάζει όλους τους τομείς. Ε, πρέπει να σας πω λοιπόν το εξής. Αποκόμισα την εντύπωση ότι ε, είσαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σήμερα βέβαια μιλάμε για τον προεπλογισμό του 2012. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες ε, πολύ σημαντικές ε, συζητήσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα σενάρια. Ας πούμε, ο συνάδελφος κ. Φέρμη αναφέρθηκε στις εργασίες της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Εργασίες που είναι πολύ σημαντικές. Ή αν θέλετε η συμμετοχή των κρατών μελών. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ πολύ ένας, ε, ένας σημαντικός στόχος για να ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός του 2012. Πρόκειται λοιπόν για έναν προϋπολογισμό ο οποίος ε, ε, οφείλει να λάβει υπόψη τις εργασίες ΣΟΥΡΕ. Το περιθώριο βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό ε, και το θέμα που τίθεται είναι να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Γι' αυτό λοιπόν καλώ τους ε, συναδέλφους να είναι ρεαλιστές, να είναι πολύ συγκεκριμένοι, να ε, ξεκινήσουν ήδη με τα πρώτα πιλωτικά προγράμματα και σας καλώ πρώτα απ' όλα να αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία στις αναλύσεις ε, που υπάρχουν σχετικά με τα περιθώρια. Γιατί τα περιθώρια για αυτές τις δράσεις ε, είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Ε, τα περιθώρια είναι πραγματικά πολύ μικρά. Ελπίζω λοιπόν ότι το θέμα του προϋπολογισμού θα είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει ιδιαίτερα την Επιτροπή σας και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και θέλω να πιστεύω ότι ευθύ εξ αρχής θα οριστούν οι ε, προτεραιότητες για το 2012 έτσι ώστε τελικά ε, να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο σε πιλωτικά προγράμματα και σε άλλα βέβαια. Ε, θα χρειαστεί ίσως να γίνουν και κάποιες αλλαγές στους αριθμούς. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι ακόμα δεν έχουν οριστεί τα κονδύλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μετά τη συζήτηση που κάναμε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς πολυμερείς οργανισμούς, συνεχίζουμε τη σημερινή συνεδρίαση με ένα παρεμφερές θέμα, που είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο με θέμα την επόμενη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο συγγητής έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο σύστασης, το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει στην ομάδα εργασίας για τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένα Έθνη και μέσα στο λόγο στον συγγητή μας για να συνοψίσει τη βασική του σύσταση. Κύριε Λάμπστορφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς όπως πολύ σωστά είπατε, στην ομάδα εργασίας για τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε συζητήσει μια φορά την έκθεσή μας Τώρα ε, πρέπει να κάνουμε μια τεχνική προσαρμογή γιατί ε, για λόγους διοικητικού χρειάστηκε λίγο να συντομεύσουμε το κείμενο, δεν αλλάζει όμως τίποτα στην ουσία. Ε, για εκείνους τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία αυτή, πρόκειται για μια σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες που έχουμε στα Ηνωμένα Έθνη στην 66η Σύνοδο της ε, Γενικής Συνέλευσης ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έρχεται να ε, βασιστεί στα προηγούμενα χρόνια σε μια ε, αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη. Ήρθαμε σε επαφή με τους εταίρους μας εκεί, με τους συνομιλητές μας για να ακούσουμε ποιες είναι οι ανάγκες τους, ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. Είναι μια πάγια συνάντηση και επίσκεψη που κάνουμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε διάλογο με ε, τα κράτη-μέλη, με τις αντιπροσωπείες, τώρα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με διάφορα προγράμματα ε, του ΟΗΕ και τα λοιπά. Äh το πόσο σημαντικά είναι τα Ηνωμένα Έθνη δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Είδαμε ε, πρόσφατα τι συνέβη με το ψήφισμα 1973 είναι πολύ αποφασιστικά. Οι προτεραιότητες της έκθεσης μου όμως ε, δεν είναι στα πλαίσια της επικαιρότητα. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας οργανισμός μεγάλος, περίπλοκος, με πολλές προκλήσεις. Ποιες είναι οι φετινές προτεραιότητες. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η εκτελεστική μας εξουσία πώς ασκεί το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Εθνών, πώς τη διαμορφώνει και πώς την αντιλαμβάνεται. Ε, ε, η οικοδόμηση της ειρήνης, peace building, στα γερμανικά δεν υπάρχει καμιά λογική έκφραση, και διαχείριση της κρίσης και ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτά τα τρία θέματα κάνουμε συστάσεις. Υπάρχουν και κάποια άλλα κεφάλαια στο σχέδιο έκθεσης που είναι πιο σύντομα για τους εξής δύο λόγους. Τον πρώτο σας τον είπα προηγουμένως ε, γιατί έχουμε περιορισμούς χώρου, το ένα και το δεύτερο συνειδητά το θέμα της αναπτυξιακής συνεργασίας που είναι σημαντικό ε, το έχουμε κρατήσει σε μικρά πλαίσια γιατί είναι παραδοσιακή η καλή συνεργασία μας με την Επιτροπή Ανάπτυξης και θέλουμε να συνεχιστεί και φέτος και περιμένουμε γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης για να τη συμπεριλάβουμε στο έγγραφό μας. Έρχομαι στο πρώτο σημείο, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι εδώ ο κύριος Γκυμαράες, βέβαια δικιά του δουλειά είναι, ε, δεν είναι εύκολη και δεν σας ζηλεύουμε καθόλου, ε, γιατί στην αρχή, στην πρώτη απόπειρα, ε, η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης αντέδρασε κάπως στεναρά. Εμείς θέλουμε μεγάλη συμμετοχή, ε, να έχουμε επιρροή, ε, αντίκτυπο, να φαινόμαστε εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα τονιστεί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στη Γενική Συνέλευση. Ε, δικαίωμα ομιλίας και ε, υποβολής προτάσεων και της ΥΠΑ της εκπροσώπου και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Γενική Συνέλευση. Ε, η κατάσταση είναι καλύτερη λίγο στο Συμβούλιο Ασφαλείας από τη Γενική Συνέλευση. Το δεύτερο αφορά την ασφάλεια και την ειρήνη. Είναι λίγο πιο επιχειρησιακή η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για την προστασία και την ευθύνη που έχουμε να προστατεύουμε. Στην ομάδα εργασίας διαπιστώσαμε ότι ε, θα πρέπει το στοιχείο αυτό να τονιστεί περισσότερο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαν αυτό το αποτέλεσμα οι συζητήσει στην ομάδα εργασία, διότι ε, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία τη 26η Φεβρουαρίου για τη Λιβύη, όχι το τελευταίο τώρα, το προηγούμενο, ε, για πρώτη φορά αναφέρει την ευθύνη προστασίας, responsibility to protect. Για πρώτη φορά αυτή η έννοια αποκρισταλώνεται σε επίσημη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, ε, σε σχέση με μια τρέχουσα και επίκαιρη κρίση. Αυτό σημαίνει ότι θα μπει τελικά ως κανόνας και διάταξη στο διεθνές δίκαιο αυτό, υποχρέωση που έχουν οι Διεθνή κοινότητα να προστατεύει ε, τον πληθυσμό. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό. Το δεύτερο σημείο, λοιπόν, κεφάλαιο που είναι σημαντικό στην ασφάλεια και στην ε, ειρήνη είναι μια ευρεία στρατηγική οικοδόμηση ασφαλείας και με αναπτυξιακά στοιχεία. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη, καλύτερη συνεργασία της ειρηνευτικής δύναμης και της διατήρησης της ειρήνης, το peace building και το peace keeping. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό το βήμα και αποφασιστική σημασία έχει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αποστολή ειρηνευτική μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας, όχι τόσο τη διατήρηση ειρήνης. Όποιος γνωρίζει τα Ηνωμένα Έθνη ξέρει ότι καμιά φορά γκρινιάζουμε για τα προβλήματα που έχουμε να ψηφίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεννοηθούμε. Στα Ηνωμένα Έθνη τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Ακριβώς αυτό το σημείο θα επιθυμούσα, ακριβώ, επειδή είναι τόσο μεγάλη η καινοτομία και ο νεοτερισμός, να πετύχει. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους άλλους, έχει σημασία ε, να βελτιωθεί ο συντονισμό με διαφόρους περιφερειακούς εταίρους. Αυτό ισχύει και για τη διαχείριση κρίσης. Ε, ας πούμε, η συνεργασία Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης ε, με υποπεριφερειακούς οργανισμούς επίσης θα πρέπει να συζητούμε. Μόλις επιστρέφω από την Γουινέα και είναι πολύ ενθαρρυντικέ οι εξελίξει και είχα πολύ θετικέ εμπειρίε με την υποπεριφερειακή οργάνωση εκεί. Ε, τώρα, για τον αφοπλισμό και ιδιαίτερα τον πυρηνικό, Το 2010 ε, είχαμε τη διάσκεψη που ήλεγχε το πώς εφαρμόζεται η ε, συνθήκη μη διάδοσης και τώρα έχουμε και τα συμπεράσματα και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας συνεισέφεραν πάρα πολύ επικοδομητικά και τα έχω βάλει στο κείμενο. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τώρα είναι μερικά θεσμικά ζητήματα. Παράδειγμα, και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, πώς θα συμπεριλαμβάνω αυτά, τι γίνεται με το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, πώς λέγεται, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, πώς βελτιώνεται η ε, εξουσία του και οι αρμοδιότητες του, αλλά και ε, η ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, για να το πω απλά, πέταξε έξω από αυτό το Συμβούλιο τη Λιβύη από τότε που άρχισε ο κύριος Καντάφη να πυροβολεί τον πληθυσμό του. Και νομίζω θα ήταν πολύ πιο λογικό να μην δεχτούμε καν στους κόλπους αυτής της Επιτροπής ε, από την αρχή τη Λιβύη, όχι να την πετάμε έτσι έξω. Ε, αυτά λοιπόν, τη διαδικασία επιλογής για το ποιο συμμετέχει και έχει σημασία. Άλλο, κατάργηση ανατικής ποινής, τώρα έχουμε ένα δικαιοστάσιο ε, το θέμα καταπολέμησης των βασανιστήριων, δικαιώματα των παιδιών, θρησκευτικά δικαιώματα και ε, δικαιώματα των γυναικών. Με χαρά να απαντήσω και άλλες ερωτήσεις όταν μπούμε στη συζήτηση, ιδιαίτερα τις σχέσεις των Ηνωμένων Εθνών με τις λεγόμενες ε, ε ομάδες G g G7, G8, G20. με χαρά να απαντήσω λοιπόν σε ερωτήσεις των συναδέλφων και περιμένω τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Ευχαριστούμε, ο κύριος Πρέντα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπσντορφ για την τόσο παραγωγική πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε για το σχέδιο του κυρίου Λάμστορφ, ο οποίος ε, είχε την ευγένεια να συμπεριλάβει κάποιες από τις ε, προτάσεις μου. Θα ήθελα παρόλα αυτά να υποβάλω κάποιες ε, άλλες τροπολογίες και θα ήθελα να σχολιάσω δύο-τρία εξαιρετικά σημαντικά κατά με ζητήματα. Πρώτον, θα έπρεπε να αναφερθούμε στο εξής. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιώντας το ίδιο μήνυμα για όλους αλλά που θα ακούγεται από διάφορες φωνές Μόλις έχουν τοποθετηθεί και εκφράσει την ε, άποψή τους ε, τα κράτη-μέλη, ε, μπορεί να αναβαθμιστεί το ειδικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το ότι υπάρχουν πολλά κράτη που ανήκουν στα, στα Ηνωμένα Έθνη. Σχετικά τώρα με το, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το δικαίωμα ψήφου, ε, θα πρέπει να επιδιώξουμε μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, οι περιφερειακές ε, ομάδες έχουν το δικαίωμα ψήφου και οι... προτείνονται κάποιοι υποψήφοι στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα χρειάζεται συντονισμός για να προτείνουμε τους σωστούς υποψηφίους ε, σε αυτό το Συμβούλιο. Επίσης θα έπρεπε να λύσουμε το πρόβλημα του διευρυνόμενου χάσματος ε, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου στην Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πέραν αυτού, ε, θα μπορούσαμε να πούμε στο σχέδιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, συνδράμει με άνω του 38% στον προϋπολογισμό του, των Ηνωμένων Εθνών. Άρα φέρει και μεγάλη ευθύνη. Θα υποβάλω και άλλες τροπολογίες, πάντως συγχαίρω τον εισηγήτη. Ευχαριστώ κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρε Λάμπστορφ το είχαμε πει και στην ομάδα εργασία, είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, είναι πολύ καλή η δουλειά του. Και εγώ θεωρώ ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει πρωταγωνιστή στην παγκόσμια πολιτική και αυτό να φαίνεται και στον ΟΗΕ. Υποστηρίζω πλήρω αυτές τι παραγράφου. Θα πρέπει να καταφέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γενική Συνέλευση ε, και μίλησε και για το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Αλεξάνδρ Λάνσορφ να ε, κάνει τη φωνή της να ακούγεται, εν πάση περιπτώσει. Ε, αυτό που θα ήταν χρήσιμο ήταν μια καλύτερη διασύνδεση, έτσι, μια καλύτερη και πιο αρμονική διασύνδεση των θεσμικών οργάνων των Βρυξελών με την αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη. Αυτό δεν συνέβη στο κείμενο για τη Λιβύη. Ε, πήγε στραβά, απέτυχε το πείραμα γιατί οι ε, χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μίλησαν με την ίδια φωνή. Και το G8 και το G20 έχουν έκτακτα όργανα, ειδικά που έχουν και αυτό το ρόλο του. Σωστό είναι αυτό. Θα πρέπει όμως να πιέσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον όχι, διορθώνει ο μιλητή, ο ΙΕ να παραμείνει ε, το κεντρικό ε, όργανο για την παγκόσμια συνεργασία και θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία των συζητήσεων του G8, του G20 με ε, τον ΟΗΕ. Για τη στρατηγική ειρήνευση γνωρίζουμε ότι η φτώχεια και η καταστροφή του περιβάλλοντος πολύ συχνά οδηγούν σε πολέμους. Είναι ενιαία λοιπόν αυτή η αντίληψη και θα πρέπει να την ε, τονίσουμε. Να έχουμε μια πολιτική πιο συντονισμένη της παγκόσμιας κρίσης. για να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε τις κρίσεις αναπτυξιακή πολιτική, προστασία του περιβάλλοντος και τέτοια ε, στοιχεία. Στην έκθεση αυτή ε, έχουμε έκτακτο ειδικό κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρικανική Ένωση και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, είναι η γειτονική μας Ήπειρος και δεδομένων των γεγονότων στη Βόρεια Αφρική θα μπορούσε κανείς να προσθέσει ακόμα κάτι. Η Βόρεια Αφρική θα πρέπει να απασχολεί όλο και περισσότερο τον ΟΗΕ πλέον και από κοινού και χωριστά ε, θα πρέπει να κάνουμε συμπληρωματικές τροπολογίες. Τώρα, κατά πολέμηση τρομοκρατίας. Βεβαίως παραμένει μέγα ζήτημα και αυτό και τονίζεται ιδιαίτερα συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εντάξει, σαφές είναι αυτό. Γιατί όχι και με τη Ρωσία, γιατί σε πολλές ε, χώρες υπάρχουν προβλήματα ε, τρομοκρατίας. Είτε θα κατονομάσουμε ε, περισσότερες της μιας χώρας είτε κανέναν, γιατί δεν έχει ε, απόλυτο νόημα. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος κοίταξα το θέμα της προστασίας του κλίματος. Περνάμε από την COP16 στην COP17 πλέον. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πολιτική στα πλαίσια των, της σύμβασης ε, του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ε, εξακολουθεί να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε ούτε να αδρανίσουμε και ο, ο, δικός χάρτης για το 2050 που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δείχνει το δρόμο, μας προσανατολίζει για το πού θα πρέπει να πορευθούμε και ίσως θα μπορούσαμε να του συμπεριλάβουμε. Θα είμαι σύντομος λοιπόν. Αλεξάνδρ Λάμστορφ, εγώ νόμιζα ότι θα έπρεπε να αναφέρουμε και πάλι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, να το ενισχύσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το όργανο και είναι πολύ ενδιαφέρον που για πρώτη φορά συμμετείχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έκλειση ε, προς το Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο ε, πολεμούσαν εδώ και χρόνια. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ακόμα να διευρυνθεί η εντολή του Διεθνούς ε, ποινικού δικαστηριού γιατί έχω υπόψη μου τεράστια εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος ε, ε, στον κόσμο όπου δεν μπορεί κανείς να προσφύγει πουθενά. Αυτό είναι ένα κενό στην παγκόσμια ένωμη τάξη. Ορισμένοι ζητούν και οι Ιταλοί νομίζω ζήτησαν ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ποινικό δικαστήριο. Δεν ξέρω κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο. Τελειώνω. Ο Αλεξάνδρ ως τελευταίο σημείο, είπε ότι ε, ε, θα πρέπει να ε, συμμετέχει περισσότερο το κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά, έχει οριμάσει ο χρόνος να συμμετέχουν. συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών, αλλά το σώμα που εκπροσωπεί τους πολίτες, το κοινοβούλιο όχι. Και εγώ θα το συμπλήρωνω αυτό ότι ε, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου για μένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ ασαφής. Και στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε ένα όργανο ε, στο σύστημα του ΟΗΕ όπου να εκπροσωπούνται τα κοινοβούλια. Το, η IPU, η Διεθνής Κοινοβουλευτική Ένωση, είναι παρατηρητής, εντάξει, αλλά ε, τα κοινοβούλια παρατηρητές είναι πραγματικά. Δηλαδή, ισοδυναικέ για μένα αυτό δεν έχει κανένα αντικείμενο. Τι να το κάνω το καθεστώ του παρατηρητού. Δεν ε, ε, ε, ανταποκρίνεται σε εκλεγμένα κοινοβούλια τον κόσμο και θα κάνω και μια τροπολογία μαζί με άλλους, αν μη τι άλλο να αρχίσει αυτή η συζήτηση για μια κοινοβουλευτική συνέλευση στα πλαίσια του συστήματος του ΟΗΕ, αντίστοιχα με την κοινοβουλευτική συνέλευση στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε που μετά από δεκαετίες εξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε την έκθεση ε, και θα κάνουμε και κάποιες συμπληρωματικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Merci. Euh, euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Λαμπστρόφ. Είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση που θα την ψηφίσουμε και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν ήδη σε σχέση με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συστήματος των ΗΕ. Εθνών. Εγώ θα περιστώ σε ορισμένα θέματα για τα οποία θα καταθέσουμε και τροπολογίες. Όσον αφορά το θέμα του πυρηνικού αφοπλισμού, στο σημείο L, εκεί με λίγα ε, λόγια αναφέρεται τι ακριβώς ε, πρέπει να συμβεί ε, και νομίζω εκεί λέμε με απόλυτη σαφήνεια ότι ε, θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα πιο γρήγορο αφοπλισμό, ποινικό αφοπλισμό με πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Δεν θα αναφερθώ βέβαια σε συγκεκριμένη διατύπωση. Όσον αφορά τώρα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, εκεί ενδέχεται να έχουμε διαφορετική άποψη, γιατί κυρίως το ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο αρχή Σωστό είναι αυτό, όμως είναι σε αντίφαση με το σημείο F όπου λέμε ότι ε, στηρίζουμε τις ε, προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Αυτά βέβαια πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με την εφαρμογή και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακούσαμε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων ε, Πολιτειών ότι θα συνεχίσει όμως να συλλαμβάνει υπόπτους και να μην αναφέρεται πού ακριβώς ε, θα κρατούνται οι ύποπτοι αυτοί. Αυτό είναι αντίφαση. Επίσης, ε, στην παράγραφο αυτή θα προτείνουμε να σκεφτούμε το κατά πόσον θα πρέπει να αξιολογούνται αυτοί οι κατάλογοι των τρομοκρατών. Γιατί δεν είναι ε, σαφές το πώς συντάσσονται οι κατάλογοι. Ούτε ξέρουμε ποιος μπαίνει στο κατάλογο, ούτε και ποιος βγαίνει. Αυτό λοιπόν που ε, πρέπει να πούμε είναι ότι τελικά αυτοί οι κατάλογοι δεν βοήθησαν καθόλου στο να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία. Ε, από ό,τι κατάλαβα είπατε ότι κάνατε περικοπές και αυτό είναι δύσκολο κυρίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα ε, και μία προσθήκη. Ε, συγκεκριμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα στο ΕΡ. Εκεί αναφέρεται τον κατάλογο των ε, βασανιστήριων μόνο ως ένα σημείο. Εγώ όμως θα έλεγα να το διευρύνουμε όπως συνέβη και πέρυσι στο ψήφισμα όπου καλούνται τα κράτη να υπογράψουν αυτό το ε, πρωτόκολλο προσθήκη στη Σύμβαση για την κατάργηση των βασανιστήριων. Ε, δεν έχει υπογραφεί το σημείο αυτό από ε, όλα τα κράτη όπως θα έπρεπε να συμβαίνει στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει και μία παραπομπή να γίνεται αναφορά στους πρόσφυγες λόγω κλιματο, κλιματικών συνθήκων. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε να υπάρξει μία ειδική σύμβαση για το θέμα αυτό και ίσως θα μπορούσαμε να δούμε πώς το διεθνές δίκαιο μπορεί ε, να αναφέρεται στο θέμα των προσφύγων. Σας λέω λοιπόν ότι ε, αυτό θα το προσθέσουμε στην παράγραφο που αναφέρεται στις, ε, στην κλιματική αλλαγή και στις τελικές συστάσεις η διαπίστωση ότι πρέπει να γίνει συζήτηση για το ρόλο των ε, κοινοβουλίων ε, στο πλαίσιο των ΗΕ. Αυτό το βρίσκω ικανοποιητικό, ε, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρί, υπάρχει και διάσταση απόψεων. Δεν θα έλεγα ότι στο σημείο αυτό πρέπει να δεσμευτούμε σε μια συγκεκριμένη μορφή της συμμετοχής των κοινοβουλίων. Ευχαριστώ κύριος Μιγιάν Μόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Κόμι Λάνσορφ για την έκθεσή του. Είναι πάρα πολύ πλήρης και επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφερθεί κανείς σε ένα τόσο ευρύ θέμα ε, για τα Ηνωμένα Έθνη με αυτό τον κορσέ που έχουμε από τη διαδικασία και ε, κάθε φορά καλείται να επιλέξει ισορροπίες ο κάθε εισηγητής για να ε, σεβαστεί αυτά τα τόσο αυστηρά όρια και τους περιορισμούς ε, συγγνώμη για την επανάληψη. Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει, είπαμε, στην ομάδα εργασίας για το Ηνωμένα Έθνη. Θα ήθελα όμως να κάνω και μερικά σχόλια εδώ, πάρα πολύ σύντομα. Ο κύριος Λάμσοφ το γνωρίζει. Εγώ θα προτιμούσα η αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στην προσθήκη νέων μελών ε, να μην μπει στις λεπτομέρειες αν θα πρέπει να είναι μόνιμα ή μη ε, τα μέλη αυτά ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επίσης γίνεται και αναφορά σε μέλη ή μη μόνιμα. Δεν χρειάζεται το Κοινοβούλιο μπαίνει σε τέτοιες λεπτομέρειες εσωτερικής λειτουργίας του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναφέρουμε για την τρομοκρατία της Ηνωμένε Πολιτείε. Συνεργαζόμαστε σε πολλά θέματα με τις Ηνωμένε Πολιτείε, αν και διαφωνούμε κάπου για το θέμα της τρομοκρατίας. Αλλά κάπου να αναφέρουμε ότι ε, έχουν αποτελματωθεί οι συζητήσεις και πραγματεύσεις εδώ και χρόνια για τη 13η σύμβαση ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτή την παγκόσμια σύμβαση πρέπει να την ε, συμφωνήσουμε κάποια στιγμή. Κάτι τώρα που είναι λεπτομέρεια. Η ευθύνη για την προστασία στη σελίδα 6 για τη Λιβύη αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ε, τα ψηφίσματα 1970 και 1973. Δεν τα βλέπω πουθενά εγώ στη σελίδα αυτή, τουλάχιστον στο δικό μου κείμενο. Στη συνέχεια, μια μικρή λεπτομέρεια. Γίνεται λόγος ότι δεν θα πρέπει ε, να δίνεται μεγάλη έμφαση ε, στις εσωτερικές διαβουλεύσεις στα κράτη-μέλη. Αυτό χωράει παρερμηνία. Είναι πολύ σημαντικό μεταξύ των κρατομελών και στο εσωτερικό των κρατομελών να γίνονται τέτοιες διαβουλεύσεις. Εγώ δεν θα έστελνα τέτοιο μήνυμα ότι δεν πρέπει να εθαρρύνουμε. Πώς το λέτε. Ε, αναφέρομαι συγκεκριμένα στο σημείο 1α. Μείωση της έμφασης που δίνεται σε εσωτερικές διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινοτικά θέματα. Όχι, θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ε, νομίζω ότι συμφωνεί και ο κύριος Λάμστροφ. Γιατί το τελευταίο ψήφισμα, αυτό το 1973, έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των τεσσάρων κρατών μελών που αυτή τη στιγμή είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και βεβαίως να διατηρούνται ε, οι εσωτερικές διαβουλεύσεις. Κάτι άλλο επίσης λεπτομέρεια. Γίνεται λόγος για τον ΟΗΕ ότι είναι το μόνο θεμητό παγκόσμιο όργανο για παγκόσμια δράση. Εντάξει, είναι θεμητό, αλλά είναι το μόνο το μόνο που νομιμοποιείται. Οπότε κατά αναλογία το G8 και το G20 δεν είναι ε, θεμητά. Μπορεί να είναι άτυπα όργανα, αλλά δεν θα έλεγα αθέμητα. Εγώ δεν θα βάζα το όλοι ότι είναι ο μόνος ε, ε, νόμιμος οργανισμός, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει και πάλι σε παρερμηνίες, ότι άλλοι δεν είναι νόμιμοι. Είναι υπερβολικό αυτό. Και η ε, αναφορά στην Αφρικανική Ένωση, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, εγώ θα βάζα και τον Αραβικό Σύνδεσμο, που είναι πάρα πολύ της μόδας ως περιφερειακός οργανισμός. Γιατί μόνο ε, η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας κουράσω και ε, ε, να μακρηγορήσω. Θα κάνω κάποιες μικρές τροπολογίες. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Ξέρω πόσο δύσκολη η δουλειά του, δεδομένων των διαδικασιών και των διοικητικών περιορισμών για τις εκθέσεις μας. Ευχαριστώ. Ε, ενημερωτικά μόνο, λέει ο Πρόεδρο. η συζήτηση που είχε προβλεφθεί για την Τουρκία δεν θα λάβει χώρα, διότι κολλείεται η κυρία Φλότρο για λόγους ανεξαρτήτους της ε, βολήσεώς της. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μουνιές. Θέλω πολύ σύντομα να συγχαρώ τον κύριο Λάμστορφ για τις συστάσεις του. Ε, άλλη μια φορά είναι πάρα πολύ πλήρης και επιπλέον αφορά και τη διεθνή ε, επικαιρότητα που δεν είναι πάντα εύκολο να αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά θέματα που θέλω να περιλαμβάνει το σύστημα. Και ε, η σχέση ανδρών και γυναικών, νομίζω θα πρέπει να γίνεται κάποια αναφορά ε, και στις γυναίκες στη δομή των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης θα πρέπει να γίνει κάποια αναφορά και στο τέλος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως ε, στοιχείο ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών ε, οργανισμών και νέα πηγή εισοδημάτων και πόρων. Γιατί είναι και στη συζήτηση για την παγκόσμια διακυβέρνηση και η ειρήνευση, το peace building που αναφέρει και ο Σλάμστροφ και το όργανο και το μέσο σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να σκεφτούμε τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με τον πυλώνα που αναφέρεται στην οικοδόμηση της ειρήνης. Μήπως το αφήνουμε λίγο ε, απογυμνωμένο, αν όχι από αρμοδιότητες, αλλά από πόρους, από προσωπικό και από κοινοτικά ε, στοιχεία. Θα ήθελα μόνο να φέρω αυτά τα θέματα, αλλά η έκθεση, εν πάση περιπτώσει, είναι εξαιρετική. Και ε, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα που ε, άκουσα την έκθεση και τη διάβασα στα αγγλικά και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που καμία πολιτική ομάδα δεν είχε καμία αντίρρηση, καμία ένσταση που είναι στα αγγλικά η έκθεση. Ε, καμιά φορά καταλαβαίνουμε ότι έχουμε περιορισμούς ε, από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και επιβάλλονται ορισμένε καταστάσεις για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των πραγμάτων. Δεν επειδή το αποφασίζουν οι εισηγητές. Χαίρομαι αυτή τη φορά που είναι μόνο στα αγγλικά η έκθεση, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Έτσι θα πρέπει να λειτουργεί η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πάρα πολύ έκθεση του κυρίου Λάμστροφ. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβω όλα όσα λέχτησαν. Θα εξοικονομήσουμε και χρόνο. Για μένα υπάρχει ένα θέμα που είναι σημαντικό και αφορά στην καταπολέμηση της διεθνούς ε, τρομοκρατίας. συνάδελφο Λόχπίλα είπε ότι δεν πρέπει να αναφέρονται μεμονωμένα χώρες. Εγώ θα συμπεριλάμβανα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετό καιρό μας κάνουν μάθημα ε, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η διεθνή δημοκρατία. Καμιά φορά αυτό είναι σωστό, άλλες πάλι όμως ε, όχι, σαφώς όχι. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές παραβιάζουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα άφηνα λοιπόν εκτός τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία κάθε άλλο. Βλέπω βλέπουμε ότι συνάπτονται όλο και περισσότερες διμερείς συμφωνίες για ε, θέματα ασφαλείας ε, στις αεροπορικές μεταφορές ή για τη μεταφορά τραπεζικών δεδομένων. Κάποια στιγμή κάνει χάνει κανείς τον έλεγχο. Έτσι λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι, ε, ειδικά όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, να έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα που να ισχύσει ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι εδώ δεν θα γράψουμε βιβλίο, θα πρέπει να είμαστε σαφείς, ε, περιεκτικοί, όλα να είναι κατανοητά ε, προς τα έξω και δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε τα πάντα και την τελευταία ανθιπολεπτομέρεια, να περιοριστούμε στα βασικά και ουσιαστικά. Ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης ε, και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Λάμστορφ για τη δουλειά που μας παρουσίασε πάρα πολύ σύντομα. Ε, θέλω να πω αυτά που ήδη είπε η κυρία Λοχπίλε σχετικά με τους πρόσφυγες για κλιματικούς λόγους κλιματικής αλλαγής. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε ξεχωριστά, ε, διότι δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Έχουν και αυτοί δικαιώματα. σε μία συνεδρίαση της υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρομαι ότι πράγματι θα πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας τους ε, κλιματικούς όπως αναφέρονται πρόσφυγες. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο κομμάτι της έκθεσης του κυρίου Λάμστορφ εκεί όπου αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή. Είναι λοιπόν ε, σαφές ε, ότι πρέπει στο επίκεντρο της συζήτησης, στον πυρήνα της, να αναφερθούμε και σε αυτό που ονομάζουμε κλιματική δικαιοσύνη. Υπάρχει η δήλωση του Μπαλή Common Differentiated ε, Responsibility. Αυτό πρέπει λοιπόν να το βάλουμε στον πυρήνα των συζητήσεων, γιατί αν δεν το κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, διεθνούς πειθαρχίας ε, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η τελευταία πρόταση της Κομισιόν σχετικά με το χάρτη του 2050, δηλαδή το 2050 να έχουμε μια κοινωνία χωρίς ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αυτή η πρόταση δείχνει πώς μπορούμε να περάσουμε από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς μπορούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο του ε, θερμοκηπίου κατά 80 μέχρι και 95%. Αυτά αναφέρονται όλα στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως αυτά δείχνουν ότι δεν μπορούμε να τα πράξουμε μόνοι μας. Το θέμα τους, ε, ακόμα και αν επιβληθεί η δημοπρασία των ε, εκπομπών, των ποσοστώσεων εκπομπών. παρόλα αυτά το πρωτόκολλο του Κιώτο τίθεται να αμφιβόλο. Γι' αυτό λοιπόν ας υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντλήσουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ίσως λοιπόν, αντί το σύστημα ανταλλαγής ε, ποσοστώσεων ε, εκπομπών, ανταυτού θα μπορούσαμε ίσως ε, να επιβάλλουμε φόρο διοξιδίου του άνθρακα και να επιβάλλουμε μέτρα σε εκείνους που δεν πειθαρχούν. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να είναι σαφές ότι αν τελικά υπάρξει μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, η μεταρρύθμιση αυτή να συνδυαστεί και με τη Γενική Συνέλευση εκεί ε, θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται και τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεκινήσουμε μια σοβαρή συζήτηση για τον ε, εκδημοκρατισμό αυτών των διεθνών οργανισμών. Βεβαίως οι ομάδες G20 και G8 κάτω από αυτό το πρίσμα δεν μπορούν παρά να είναι μόνο ομάδες ανάληψης ε, πρωτοβουλίας οι οποίες θα τροφοδοτούν τη συζήτηση που θα διεξάγεται στους διεθνείς οργανισμούς. Στους διάφορους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, euh, monsieur Ευχαριστούμε κύριε Γκυμαρές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίζω τη συστάση στο σχέδιο συστάσεων του Συμβουλίου για την 66η Γενική Συνέλευση. Η ομάδα εργασίας για αυτό το θέμα άρχισε να εργάζεται και φυσικά θα ε, βοηθηθεί τα μάλλα από τις συστάσεις αυτές. Ε, τον ε, Απρίλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει διάφορα σοβαρά ζητήματα ο κύριος Λάμστορφ και φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε, συνεχίσουμε το διάλογο. Δύσκολα μπορώ να σας πω ε, Ποιε θα είναι οι προτεραιότητε ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ε, όπως θα παρουσιαστούν ε, στην 66η Γενική Συνέλευση. Εμεί θα θέλαμε ένα πιο συνοπτικό κείμενο, να έχουμε συγκεκριμένε προτάσει που θα συνδέονται με τι τρέχουσε εξελίξει, τι μελλοντικέ εξελίξει και να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Πέρυσι κατορθώσαμε να περιορίσουμε, να περιστήλουμε το περιεχόμενο του κειμένου και νομίζω ότι και φέτος θα τα καταφέρουμε. Πάντως, η θέση μας ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις συστάσεις σχετικά ε, με τους τρεις πυλώνες ε, του ΟΗΕ, δηλαδή ε, ειρήνη, ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα επιδιώκουμε μεγαλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη συνέπεια στις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κόλπους του ΟΗΕ. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να ε, υπερψηφιστεί το σχέδιό μας ε, στη Γενική Συνέλευση ε, ούτω ώστε να μπορέσει να παρέμει στη γενική συζήτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη της Ένωσης έχει δώσει νέα όθηση σε όλη την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και φυσικά θέλουμε να συμμετάσχετε στις γενικότερε εργασίες τη Γενικής Συνέλευση. Θα, θα ήθελα επίσης να σε ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις. Έχει ληφθεί απόφαση για την επίσημη υποβολή του ψηφίσματος ε, στη Νέα Υόρκη μετά από όλες τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει, ιδιαίτερα από το Σεπτέμβριο και μετά, και από το ψήφισμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι επιδιώκουμε τη λήψη απόφασης ταυτόχρονα εξακολουθούμε ε, να δείχνουμε ότι επιδιώκουμε τη συνένεση, ενώ ούτως ή άλλω τους κόλπους ε, των Ηνωμένων Εθνών καταβάλλονται προσπάθειες για να καταλήξουν στο τελικό κείμενο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα και θα επανέλθουμε όταν επίκειται η ανάληψη δράσης ε, για το θέμα του ΟΗΕ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και για τα πολλά επικοδομητικά σχόλια και παρατηρήσεις. Πολύ χρήσιμο. Θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ τον κύριο Κιμαράες και τους υπολείπους και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Είχαμε άριστο διεύλο επικοινωνίας για όλα αυτά τα θέματα. Είναι κάτι το οποίο βελτιώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ χρήσιμο. Συγχαρητήρια για την απόφαση που πήρατε να υποβάλλετε επίσημα το σχέδιο ψηφίσματος και ελπίζω αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά. Ε, και νομίζω ότι εκφράζω και την αίσθηση συναδέλφων. Θα αναφέρω λίγα μόνο θέματα. Ε, μια πολύ γενική παρατήρηση πρώτα απ' όλα που έχει να κάνει με αυτό που είπε ο συνάδελφος πρώτη για το κλίμα. Όταν αναφέρουμε τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα εδώ, το θέμα δεν είναι τόσο πολύ για το περιεχόμενο, αλλά για το ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό. Ότι είναι ο μόνος οργανισμός που έχει αυτή την ομιμότητα του παγκοσμίου ε, ε, ρόλου για να θεσπίζει διεθνές δίκαιο. Και επίσης ε, για τις άλλες επιτροπές ε, δεν θέλω να προεξοφλήσω τη δική τους θέση. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να παραμείνει η διαδικασία κατοχυρωμένη στα Ηνωμένα Έθνη άλλα θέματα. Χαίρομαι που ε, αναφέρεται αυτό το θέμα των ανδρών και των γυναικών. Είναι καινούργια τα ε, ε, πράγματα. Θα έρθει αρμόδια εδώ πριν τη συνεδρίαση στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργασία. Ε, Επίση, ε, θα συζητηθεί στο κοινοβούλιο θέμα, θα τεθεί σε ψηφοφορία. Το θέμα τη καταπολέμηση τρομοκρατία και η διάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται κριτική γιατί αναφέρουμε ε, τις Ηνωμένες ε, γιατί εκεί έγινε η 11η Σεπτεμβρίου και φέτος έχουμε τη 10η επέτειο της 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, η κριτική ε, έχει να κάνει με την ανεπάρκεια στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και είναι ευρεία η ε, αλλά γιατί να αναφέρουμε τη Ρωσία ως ε, αντίβαρο ή αντιπαλωδέως. Η αντίπαλο, η κατασταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ χειρότερη. Για ποιο λόγο να φέρουμε τη Ρωσία ξαφνικά και να να υπενηχθούμε ότι οι ρωσικές αρχές κατά πολέμης τρομοκρατίας υπερτερούν κατά πολύ απέναντι στις αμερικανικές. Δεν ξέρω το συζητήσουμε και στην ομάδα εργασίας. Και αν αναφέρουμε Ηνωμένε Πολιτείε και Ρωσία θα πει ο άλλος γιατί δεν αναφέρει στην Ινδία. Βλέπει Βομβάη, οι Φιλιππίνες και πάει λέγοντας. Έτσι, ε, ως Ευρωπαίοι νομίζω ε, θα πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον να φέρουμε μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως είμαι πρόθυμος να το συζητήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Προφανώς, το είπε και ο Γιώ Λάινεν, θα μιλήσουμε για τα γεγονότα της Βορειοαφρικής και το ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης. Και αυτό που είπε ο Φρανσίσκο για τον Αραβικό Σύνδεσμο για την κοινοβουλευτική συνέλευση και πάλι θα γίνει ζωηρή συζήτηση και ψηφοφορία, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο συμφωνώ κατά 95% με το Γιολάινεν, για τον ΟΗΕ σε αυτό το συγκεκριμένο διαφωνώ. Νομίζω ότι είναι υπεραπλουστευτικό να λέμε ότι ας κάνουμε δημοκρατικά τα Ηνωμένα Έθνη, ε, προσκαλώντας βουλευτές από όλο τον κόσμο στη Νέα Υόρκη. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα συνεδριάζουμε μαζί με κάποιους από την Κινέζικη, από τη Βορειοκορεατική Βουλή ας πούμε ή τη Βουλή της Κούβας και αυτό υπό το μανδύα της Δημοκρατίας. Να γίνει αυτή η συζήτηση, τα είπε και η Μπάρμπαρα Πίλερ. μπορεί να υπάρχουν σωστοί τρόποι να προχωρήσουμε που δεν τους έχουμε σκεφτεί ακόμα, αλλά η κοινοβουλευτική συνέλευση δεν μου φαίνεται ε, η βέλτιστη λύση εμένα. Οι κλιματικοί πρόσφυγες βεβαίως θα πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή έπεσε θύμα στο βωμό της, ε, ε, του χώρου και του περιορισμού που είχα αυτό το θέμα για το ICC επίσης το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχουμε τους φίλους του Διεθνούς Δικαστηρίου ε, υπό την ηγεσία της Μπάρμπαρα Μπίλερ και ε, το Κοινοβούλιο είναι πολύ αλλά ενημερωμένο και μπορεί να τοποθετηθεί και για αυτό το θέμα. Πάντως, να σταθμίσουμε, να δούμε πώς θα μπουν αυτά. Αυτό που θέλουμε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να είναι στελεχωμένη με ε, σωστό τρόπο και σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στη Νέα Υόρκη. Το συζητήσαμε και πέρσι ε, για τον προπολογισμό ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοσιονομική ουδετερότητα σε αυτά τα θέματα ε, με ε, το άχθος που έχει φορτιστεί τώρα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και έχει αναλάβει τόσα πολλά από τις εκπεριτροπή προεδρίες. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ε, περιμένω τη συζήτηση και τη ψηφοφορία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ κύριε Λάμπστορφ. Δύο ενημερωτικά σχόλια. Προθεσμία κατάσταση απολογιων 31 31η Μαρτίου και δεύτερη ε, συζήτηση και ψήφιση στην Επιτροπή μας στις 12 Απριλίου. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Μπάσλεϊ θα έρθει που είναι επικεφαλής της νέας μονάδας ε, του ΟΗΕ για τι γυναίκε, θα έρθει στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Τούτη εδώ την Πέμπτη μεθαύριο, 24 του μηνό και θα συμμετέχει σε συνεδρίαση τη Επιτροπή Γυναικών από τι 9 μέχρι τι 10.30 και η ε, συνεδρίαση αυτή θα διευρυνθεί ε, και προς τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που επιθυμούν να λάβουν μέρος. Λήξη συνεδρίασης.